Κυρίε Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο και πέντε η ώρα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Και καλώς ορίζω θερμά όλους τους παρευρισκομένους στην ημέρα για την ε, πολιτική, για το εμπόριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε την εκδήλωση αυτή έχει βέβαια πολύ συγκεκριμένο υπόβαθρο ως Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Θέλουμε να συζητήσουμε ζητήματα νομιμότητας και ε, εγκαθίδρυσης ανάπτυξης ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε νέα πρόταση της Επιτροπής για νέα προσέγγιση στην ε, πολιτική εμπορίου, το trade for all, εμπόριο για τους πάντες. Έτσι λοιπόν, έναυσμα για αυτή την ε, ημερίδα για την ε, εμπορική πολιτική είναι να αξιολογήσουμε πάνω απ' όλα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτή η νέα πολιτική για το εμπόριο στην πράξη πώς αναπτύσσεται και τι είδους προοπτικές μπορεί να υπάρξουν για το μέλλον. Φυσικά όλα αυτά με υπόβαθρο. Την διαπίστωση για μια πολύ διαφοροποιημένη εικόνα ως προς την εμπορική πολιτική. Έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Εδώ δίπλα μου έχουμε τον εισηγητή για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο έχει βέβαια δώσει νέο φως στην συζήτηση για την εξωτερική πολιτική για το εμπόριο, αλλά βέβαια και με υπόβαθρο τις ε, λαϊκιστικές φωνές που τάσσονταν κατά του διεθνούς εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπέρ του Brexit και της εκλογής βεβαίως ενός Προέδρου στις ΗΠΑ, ο οποίος ρητά έχει ταχθεί κατά της ε, επεκτατικής, όπως την είχε χαρακτηρίσει κατά την προεκλογική του εκστρατεία, εμπορικής πολιτικής. Αυτό για πολλούς και στις χώρες μας γεννά ανησυχίες σε σχέση με την εμπορική πολιτική. Η εμπορική πολιτική λοιπόν σήμερα δεν είναι ένα μεμονωμένο κομμάτι πολιτικής. Έχει γίνει αποδεκτή πολλαπλώς ως τρόπο ζωής, αλλά ταυτόχρονα τα βρίσκεται και ενώπιον πολλαπλών προκλήσεων. Αυτά ειδωμένα μαζί και με την παγκοσμιοποίηση που έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Αν κοιτάξουμε από το 1980 μέχρι σήμερα, κυρίες και κύριοι, και κύριοι το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει πολλαπλασιαστεί. Ο παγκόσμιος εμπορικός όγκος έχει 900 ε, πλασιαστεί. Ο παγκόσμιος όγκος επενδύσεων άμεσων ξένων επενδύσεων έχει πολλαπλασιαστεί κατά λόγο 2.500. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια εκτεταμένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία η οποία τώρα εκτός από το επίπεδο στο οποίο ήμασταν παλιότερα της απλής ανταλλαγής προϊόντων τώρα έχει περάσει στο στάδιο της παραγωγής αξίας με πολύ μεγάλο όγκο πρώτων υλών στις, ανταλλαγές, στις συναλλαγές και 30% μόνο ε, προϊόντων, ολοκληρωμένων προϊόντων. Και αυτό αποδεικνύει πόσο εξαρτημένος είναι ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη από αυτές τις συναλλαγές. Όσο και να αυξάνονται οι εξαγωγές μας, είναι ταυτόχρονα εξαρτημένες και από τις εισαγωγές. που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν τα προϊόντα αυτά. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι ξεκάθαρο ότι η εξωτερική εμπορική πολιτική δεν πραγματεύεται πλέον μόνο ζητήματα τελωνιακά αλλά και προδιαγραφών, προδιαγραφών κρουσία του καταναλωτή, ανθρωπινών δικαιωμάτων, στόχων αηφορίας. Είχαμε άλλωστε τα τελευταία χρόνια και τους στόχους της αηφορίας και όλα αυτά εγγράφονται μέσα σε μια πολιτική εμπορική που θέλει να διαμορφώσει τον κόσμο στη νέα του μορφή. Όλα αυτά μέσα στην ε, αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται επιφυλακτικοί απέναντι στην παγκοσμιοποίηση γιατί θεωρούν ότι ξεφεύγει από τον έλεγχό τους η κατάσταση. Εμείς μιλούμε για προδιαγραφές και κανόνες για ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και έτσι τίθεται αυτομάτως το ερώτημα των αρμοδιοτήτων. Από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμόρφωση της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να επανεθνικοποιηθεί αυτή η εμπορική πολιτική για λόγους εξυπηρέτηση εθνικών ή περιφερειακών συμφερόντων, γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός της εμπορικής πολιτικής υπονομεύει και το, ε, την πορεία για την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να σταθμιστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, αλλά ταυτόχρονα και να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να ε, απλουστεύσουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή, τις διαδικασίες αυτές, έτσι ώστε να παράγουν ταχύτερα αποτελέσματα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητα δράσης με την ταυτόχρονη διαφύλαξη των δυνατοτήτων δημοκρατικής παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, αντιπροσωπευτικού οργάνου. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια γενικότερη συζήτηση στην κοινωνία και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε να θέσουμε και το ζήτημα της ευθύνης των εθνικών κυβερνήσεων. Αφενός με να έχουμε εμπορικές συμφωνίες με συμμετοχή και σύμπραξη ε, εθνικών κυβερνήσεων, ομόφωνα λαμβάνονται οι αποφάσεις από 28 κυβερνήσεις και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αλλά και τη στιγμή της κύρωσης καθιστούν την ε, Επιτροπή και το Κοινοβούλιο υπεύθυνα για οποιαδήποτε ε, εξέλιξη και βλέπουμε να υποχωρούν, να υποχωρεί η εικόνα των εθνικών κυβερνήσεων. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία για δημοκρατική λήψη αποφάσεων και στα κράτη-μέλη να διαφυλαχθεί, πρέπει να θέσουμε επιθετικά αυτό τον όρο στη δημόσια συζήτηση και έτσι, και ξέρουμε πολύ καλά για το πράγμα μιλούμε, απαιτείται η διαφύλαξη της διαφάνειας, για την οποία και οι δύο, τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, επανειλημμένως έχουν προβεί σε ε, προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και σε επίπεδο ε, νομοθέτη, αλλά και, σε, ε, και έναντι της κοινή γνώμης. Η σαφής λοιπόν θέση ότι θέλουμε την παγκοσμιοποίηση με προδιαγραφές, με γνώμονα τον άνθρωπο, με κανόνες, με δημοκρατικό μέσα που να μην θέτουν ένα αμφιβόλο το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με μέσα διαφάνειας, με διαφύλαξη δίκαιων όρων προς το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν νομιμότητα, νομοποίηση προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα και όσο το δυνατόν καλύτερες, καλύτερη πρόοδο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε δεν θα, πρέπει να το περιορίσουμε εδώ μέσα στο κτίριό μας αλλά και γενικότερα στην κοινωνία με το Twitter, με σχόλια που μας ε, απευθύνονται. Έχουμε φτιάξει το hashtag Trade Policy Day στο Twitter για να ε, παρακολουθήσουμε και τα σχόλια των πολιτών και να τα συμπεριλάβουμε στη συζήτησή μας. Είχαμε προγραμματίσει σε δύο τμήματα τη συζήτησή μας για σήμερα. Το πρώτο τμήμα θα ασχοληθεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης στο, στη διεθνή σκηνή. Το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθεί περισσότερο με την εσωτερική διάρθρωση και την νομιμοποίηση των εργασιών. Ο κύριος Βίγκλερ και ο υποφαινόμενος θα ε, ε, προεδρεύσουμε στα δύο αυτά τμήματα και πρώτος θα αναλάβει το πρώτο τμήμα ο κύριος Βίγκλερ και το δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι και από άλλα θεσμικά όργανα. Με τους τεράστιους όγκους της παγκόσμιας οικονομίας, ε, τραπεζικών συναλλαγών κλπ. Σας λέω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου επιτρέπετε να διευθύνω την ε, σημερινή συζήτηση. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια ή δυο ομολογίες. Προέτους όταν Αρχίσαμε την οργάνωση της παρούς συνεδριάσεως, όπως είπε και ο Πρόεδρος μας, συζητούσαμε και με την Επίτροπο κυρία Μάλμστρομ, η οποία τότε μόλις είχε παρουσιάσει τη νέα ε, εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αρχική ιδέα ήταν ότι θα είναι καλό να προβούμε σε μια αξιολόγηση και σε ένα είδος feedback, ανταλλαγή απόψεων, μετά από ένα χρόνο, δηλαδή ένα έτος μετά από την παρουσίαση της ε, νέας εμπορικής στρατηγικής. Εάν ωστόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια σύγκριση, θα πρέπει να ομολογήσω ότι άλλαξε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα σε αυτό το χρόνο, από τότε δηλαδή που είχε παρουσιαστεί η νέα εμπορική στρατηγική. Και ακολουθεί τώρα η δεύτερη ομολογία μου. Λίγα λεπτά πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, συζητούσαμε με τον πρόεδρο Λάγκε, όπως ο Μπομπ Ντίλαν μόλις τώρα δέχτηκε, δέχτηκε ε, το βραβείο Νόμπελ πριν από λίγες μέρες και ανέφερε κάποιο στίχο του «Αλλάζουν οι καιροί», λέει ο στίχος αυτός «The times they are changing» και εγώ λέω ότι τώρα έχουμε πια ένα καινούριο κόσμο μπροστά μας. Αυτό είναι όλο. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι του πάνελ, η αρμοδία επίτροπος κυρία Μάλμστρομ, ο υποδιευθυντής κύριος Λάουνερ του ΠΟΕ, διευθυντής Ευρώπης του IMF, του ΔΝΤ, δηλαδή ο κύριος Φρανκς και ο διευθυντής του εμπορίου, κεφαλής διευθυντής εμπορίου του ΟΣΑ είναι επίσης παρόν. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας εδώ και θα αρχίσω αμέσως δίνοντας το λόγο στην Επίτροπο η κυρία Μάλμστρομ για να προχωρήσει στην ε, δική της παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ για την οργάνωση της συζητήσεως που είναι και πολύ επίκαιρη, ίσως και πιο επίκαιρη από τότε που στείλατε τις προσκλήσεις για να συζητήσουμε περί εμπορίου. Διότι το εμπόριο, όπως είπατε και εσείς, είναι όλο και πιο ψηλά στην προτεραιότητα των ε, όλων έχει μεγάλη αξία το εμπόριο και το αντιλαμβάνει το κόσμο αυτό. Δηλαδή φέρνει και ανάπτυξη, φέρνει και ε, ε, ευημερία. Υπάρχουν όμω και φόβοι που συνδέονται με το εμπόριο και γι' αυτό τα δύο αυτά θέματα που επιλέξατε για σήμερα, δηλαδή η διαμόρφωση τη παγκόσμια ε, εμπορική πολιτική και η νομιμοποίησή τη, είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Λίγα λόγια λοιπόν για αυτά. Χάρηκα πολύ που τελικώ μπορέσαμε να υπογράψουμε την προηγούμενη Κυριακή την συμφωνία με τον Καναδά, την συμφωνία ΣΕΤΑ και συνεργαστήκαμε στενά μαζί σας και με τους παρόντες και παρούσες ευρωβουλευτές και ελπίζω ότι θα υπάρξει υποστήριξη για τη συμφωνία αυτή, διότι η συμφωνία με τον Καναδά, η ΣΕΤΑ, είναι καλή για να μην πω, είναι καλό μάλλον, για να μην πω θαυμάσιο παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση του παγκοσμίου εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης της ίδια, διότι ο πρώτος στόχος της εμπορικής στρατηγικής είναι να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από την παγκόσμια ανάπτυξη. Και το κάνει αυτό η ΣΕΤΑ. Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς που εργάζονται στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες, στους γεωργούς. Η διαμόρφωση όμως της παγκοσμιοποίησης σημαίνει επίσης ότι πρέπει να δώσουμε την αίσθηση στους Ευρωπαίους ότι συνδιαμορφώνουν τους παγκόσμιους κανόνες. Επομένως η εμπορική πολιτική πρέπει και να προστατεύει και να προωθεί τις αξίες που υποστηρίζουμε εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνει αυτό η ΣΕΤΑ. Έχει δηλαδή διατάξεις για τα εργασιακά και τους πιο, φιλόδοξε φιλόδοξες διατάξεις από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία για την αηφόρο ανάπτυξη, προσεγγίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και διασφαλίζει ώστε Ευρωπαίοι και Καναδοί να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θέλουν να οργανώσουν τα της υγείας, της οδροδότησης και ούτω καθεξής έχει και βελτιώσει στην προστασία των επενδύσεων, που είναι τα πρώτα, για τα πρώτα βήματα για μια βελτίωση και των δημόσιων επενδύσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυτά λοιπόν όλα δίνουν μια φωνή στους Ευρωπαίους στο παγκόσμιο επίπεδο και δείχνει πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική στρατηγική και πολιτική για να διαμορφώσουμε τη μελλοντική παγκοσμιοποίηση. Trade for all, το εμπόριο για όλους όπως είπε ο κ. Βίνκλερ προηγουμένως. Θέλουμε ένα διαφανές και υπεύθυνο εμπόριο. Δεν μιλώ μόνο για τις οικονομίες. Αυτά δεν τα εφαρμόζουμε στην πράξη μέσα από την Συμφωνία ΣΕΤΑ. Προωθούμε και νέα πρόοδο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για σημαντικά ζητήματα. Και ένα από αυτά τα σημαντικά ζητήματα όπου χρειαζόμαστε παγκόσμιους κανόνες, είναι και ο ψηφιακός τομέας, ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε το δυνατόν περισσότερο από την online οικονομία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και υποστηρίζουμε και μια ε, διεθνή συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά και τη Διεθνή ε, Σύμβαση για, τα, για το Περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν φιλόδοξους και μάλιστα τους πιο φιλόδοξους στόχους στην ατζέντα μας ό,τι αφορά πολυμερείς και πλειονομερείς συμφωνίες. Έχουμε στην ΣΕΤΑ τώρα μια τελική μορφή που ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε σήμερα. Ε, σύντομα έχουμε και συμφωνία με το Βιετνάμ που προχωρεί και αυτή στην μετάφραση τώρα και αντιμετωπίζει μια από τι μεγαλύτερες προκλήσεις τη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή πώς συνδέουμε τις προσπάθειές μας με αυτές των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Και έχουμε και άλλε 20 συμφωνίε η ατζέντα μα επεκτείνεται όλο και περισσότερο και μόνο για φέτος, διότι πρόκειται για αξιολόγηση του πρώτου έτου, αρχίσαμε διαπραγματεύσει με το Μερκοσούρ, το Μεξικό, την Ινδονησία και την Τινησία. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να πράξουμε το ίδιο με την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία και Χιλή. Όπω και για την ΣΕΤΑ, όπω ισχύει για την ΣΕΤΑ, οι συμφωνίε αυτέ θα είναι οικονομικά αποδοτικέ θα αντιμετωπίζουν τους θεσμολογικούς φραγμούς, θα ανοίγουν νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις, με και επιχειρήσεις, επενδυτές και θα προσφέρουν περισσότερες ε, επιλογές στους ε, πελάτες καταναλωτές. Θέλουμε λοιπόν υψηλά νομοθετικά επίπεδα, κοινωνικά συστήματα, περιβαλλοντικά πρότυπα. Και θα είναι διαφανείς και αυτές και θα δώσουμε και φωνή στους ενδιαφερόμενους, στους stakeholders. Η πολιτική εμπορίου σημαίνει όλες αυτές τις συμφωνίες, αλλά όχι μόνον. Και βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω και για την πρότασή μας που ολοκληρώνεται σχεδόν για τα ορυκτά συγκρούσεων. Έχουμε και μια πρόταση για διατυπώσεις κατά των βασινιστήριων και επίσης για το DSP, DSP SIN για χώρες που εφόσον καλύπτουν ορισμένα ε, πρότυπα για περιβαλλοντικά δίκαια, ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω Έχουμε και εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Έχουμε λοιπόν πράγματι μια πολύ φιλόδοξη ε, παγκόσμια εμπορική ατζέντα που στηρίζει και τα ε, δικαιώματά μας αλλά και τα δικαιώματα του κόσμου. Ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα νομιμοποίησεως για όλα αυτά. Διότι όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε θα ωφελήσουν τους πολίτες μόνο εφόσον κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Ακόμη και αν υπήρξαμε πράγματι καλοί στην επίτευξη συμμονιών, πρέπει βεβαίως και να προσεγγίσουμε τους πολίτες ακόμη περισσότερο από ό,τι πριν. Ήταν καλό λοιπόν που υπογράψαμε τη ΣΕΤΑ, όμω μετά από μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Και θα χρειαστεί να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό και μέσω και βράχη πρόθεσμα για την εμπορική πολιτική, διότι ζούμε σε πολύ δύσκολου και περίπλοκου καιρού. Από τη μια μεριά το εμπόριο γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την οικονομία και την ευημερία μα από ποτέ. Πιο πολλέ εφοδιαστικέ αλυσίδε, πιο πολλέ δουλειέ, 31 εκατομμύρια, 31 εκατομμύρια ε, Θέσει εργασία στην Ένωση εξαρτώνται από τι εξαγωγέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη δουλειά, χρειαζόμαστε και περισσότερε εξαγωγέ. Η συμφωνία με την ε, Νότια Κορέα αύξησε τις εξαγωγές μας κατά 50%. Πρέπει όμω να διασφαλίσουμε κιόλας ότι θα αντιμετωπίσουμε και του φόβου που προκαλούν οι εμπορικέ συμφωνίε σε ορισμένου πολίτε. Ορισμένοι φοβούνται το ενδεχόμενο απώλεια θέσεων απασχολήσεω για λόγω του εντονότερου διεθνού ανταγωνισμού. Βεβαίω συχνά τα φορτώνουν αυτά στο εμπόριο. Το γεγονός είναι όμως ότι πολύ λίγες απώλειες θέσεων απασχολήσεως οφείλονται στο εμπόριο. Πιο πολύ είναι η αλλαγή της τεχνολογίας. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο αυτές οι θέσεις απασχολήσεως πέφτουν θύμα της παγκοσμιοποίησης. Και έχουμε βεβαίως και περιορισμούς στην δυνατότητα νομοθεσίας στο δημόσιο επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να ακούμε προσεκτικά και να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας. Να συμμετάσχουν λοιπόν οι άνθρωποι και στο εθνικό επίπεδο, τα δε εθνικά κοινοβούλια επίσης να συμμετάσχουν. Εγώ επισκέφθηκα 22 εθνικές βουλές πέρσι και θα συνεχίσω να το πράττω για να συζητήσω εμπόριο. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο διότι εσείς εκπροσωπείτε τους ε, Ευρωπαίους, είστε η διασύνδεση μεταξύ των Βρυξελών και των εκλογικών περιφερειών σας. εσεί μπορείτε να εξηγήσετε το στοιχείο της περιπλοκότητας στους ψηφοφόρους σας. Άρα ο ρόλος σας είναι σημαντικός. Και επίσης οι εθνικέ κυβερνήσει, των οποίων ο ρόλο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πολλέ από τι κυβερνήσει αυτέ, πολλοί υπουργοί, πολλέ κυβερνήσει είναι δραστηριότατοι στην διασύνδεση και στην επικοινωνία των θεμάτων αυτών με του πολίτε. Μπορούν να κάνουν ακόμα περισσότερα διότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται μια συμφωνία και την θέτει υπόψη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του κοινού, δεν είναι τότε ο χρόνο να συζητηθεί ε, η υπόθεση αυτή. Πρέπει να έχει να αρχίσει να συζητείται από τότε που δίνεται η εντολή. Άρα, είναι σημαντική η ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων για να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πώ θα αντιμετωπίσουν τι συμφωνίε και την παγκοσμιοποίηση για θέματα όπως απασχόληση, υποδομές κλπ να μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι και να παρακολουθήσουν τις, ε, την ταχύτητα των αλλαγών. Βλέπουμε λοιπόν σημαντικέ αλλαγέ στην εμπορική πολιτική, ίσως σε, σε λίγους μήνες να δούμε ακόμα πιο σημαντικέ αλλαγέ. Μπορούμε όμω με αποφασιστικότητα, ευκαμψία και ανοιχτό πνεύμα να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα και μάλιστα και να αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό που πράττουμε. Και αυτά τα πράγματα βέβαια θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων ε, σήμερα. Σα ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τι σκέψει που θέσατε υπόψη μα και τι ε, πληροφορίε, τι οποίε άλλωστε μα θέτεται συχνά τακτικά υπόψη εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά πρώτα θα υπενθυμίσω την τεράστια σημασία του ΠΟΕ στον κόσμο του εμπορίου, είτε τον παλαιό είτε τον νέο κόσμο του εμπορίου και για το γεγονός ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνεται μεγάλη συνένεση και στήριξη σχετικά με το ότι το πολυμερές σύστημα το οποίο, το οποίο οργανώνει ο ΠΟΕ πρέπει να παραμείνει ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, ανοιχτό και διαφανές. Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία και στην κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ και η δική μου αίσθηση είναι ότι η σημασία αυτή θα γίνει μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Διότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του παγκόσμιου εμπορίου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπράουνερ που είναι ε, του ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάγκε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, Επίτροπε Μάλστρομ, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σα να συμμετέχω σήμερα στην ημέρα εμπορική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λαμβάνει η χώρα σε μια στιγμή όπου το εμπόριο και οι εμπορικέ συμφωνίε όλο ιδιαίτερω κατηγορούνται από πολλού για ένα σωρό αρνητικέ ε, ε, επιπτώσεις. Αυτό έγινε σαφές στον αγώνα που δόθηκε σε σχέση με την ΣΕΤΑ και φυσικά στη διάρκεια των, ε, ε, της εκλογικής εκστρατείας των ΗΠΑ. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω την σταθερή μας δέσμευση να συνεργαστούμε με τα κοινοβούλια ώστε να προωθήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι διακυβεύεται. Ο ρόλος σας ως μέλη του Κοινοβουλίου έχει ήδη τονιστεί αυτό, είναι μεγάλη σημασία, ακόμα και σε καιρούς παγκοσμιοποίησης, όλες οι επιχειρήσεις είναι τοπικές. Πρέπει να έχετε επαφή με τους ανθρώπους των εκλογικών σας περιφερειών και άμεσα αντιμετωπίζετε τα πραγματικά αλλά και τα τεκμερώμενα ε, τις τεκμερώμενες επιπτώσεις του εμπορίου και των εμπορικών συμφωνιών. Ο ρόλος σα στην επεξήγηση των, ε, του περίπλοκου χαρακτήρα των διεθνών διαπραγματεύσεων και των υπέρ και των κατά των πολυμερών συμφωνιών είναι κρίσιμος. Η συζήτηση για το εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δύο πλευρές του κάθε επιχειρήματο. τα ωφέλη του εμπορίου και της παγκοσμιοποίηση, αλλά καθώς επίσης τις προκλήσεις που θέτουν αυτά τα δύο για πολλές περιφέρειες. Μόνο μέσω μιας ε, ενήμερη συζήτηση μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο του αθέμητου προστατευτισμού ο κόσμος ε, συγχαίει τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου και της τεχνολογικής πρόοδου. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Για 12 χρόνια ήμουν ε, το μέλος ε, που εκπροσωπούσε τη Γερμανία στην Επιτροπή για την Πολιτική Εμπορίου, την Εμπορική Πολιτική. Κάποτε ήρθα στις Βρυξέλλες με οδηγίες να αγωνιστώ ώστε να διατηρηθεί ψηλό δασμό για τις μεγάλες τηλεοπτικές συσκευές, τις μεγάλες τηλεοράσεις. Είχε μόλις δημιουργηθεί ένα νέο εργοστάσιο κοντά στο Άχεν και ο Ευρωπαίος κατασκευαστής είχε πείσει την κυβέρνησή μου ότι χρειαζόταν προστασία έναντι του ασιατικού ανταγωνισμού με τη βοήθεια ενός ε, σχετικά ψηλού δασμού. Να σας πω, αυτές οι τηλεοράσεις ήταν πραγματικά μεγάλες. Μεγάλες όχι μόνο φαρδιές αλλά και πλατιές ήταν αρκετά ε, ε, ογκώδης λόγω των τεράστιων Ε, λόγω των τεράστιων καθόδων ήταν απαραίτητε για αυτέ τι μεγάλε οθόνε. Ε, ήταν παλιά τεχνολογία. Ο κατασκευαστή είχε επενδύσει στην παλιά τεχνολογία. Είχε χάσει το τρένο τη τεχνολογική προόδου. Αυτή η επένδυση δεν μπορούσε να σωθεί ό,τι εμπορικά μέτρα και αν λαμβάναμε στην εμπορική μα πολιτική. Τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει κρατήσει ζωντανή αυτή τη γραμμή παραγωγή. Ένα άλλο παράδειγμα, ο επικεφαλής οικονομολόγος ένα Αμερικανό στον ΠΟΕ τονίζει ότι εκατομμύρια Αμερικανοί οδηγοί φορτηγών κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσει τους όταν τα φορτηγά αυτά θα αρχίσουν να καλύπτουν μακρές αποστάσεις αυτόνομα αυτό θα είναι πολύ οδυνήρο για τον κόσμο που θα, θα πληγεί. Θα πρέπει να στηριχτούν για να προσαρμοστούν. Όμως αυτή δεν είναι η εμπορική πολιτική που θα δώσει το, την εργαλειοθήκη. Η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό και δεν μπορεί ούτε και να βοηθήσει. Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτύχει η εμπορική πολιτική. Αλλά αυτό που μπορεί να επιτύχει είναι να αξιοποιήσει την, το πλήρες της δυναμικό. Έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά την πολιτική trade for all, εμπόριο για όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κινεί την εμπορική της πολιτική σε επόμενο επίπεδο μέσω των ανοιγμάτων της ε, νέας αγοράς. Ε, λυπάμαι που αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Οι συμφωνίες δεν είναι μόνο για το ελεύθερο εμπόριο. Μιλάμε, εγώ προέρχομαι από την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, όχι ελεύθερου εμπορίου. Δεν αφορά όπου ε, μόνο το ελεύθερο εμπόριο. Είναι ένα αριθμιστικό πλαίσιο που προσφέρει προβλεψιμότητα και νομική βεβαιότητα επί τη βάση των συμπεφωνημένων μεταξύ των μερών. Μεγάλα κομμάτια της δουλειά μα ε, είναι αφιερωμένα στα πρότυπα όταν πρόκειται για θέματα SPS και TBT. Οι διαδηλώσεις κατά του εμπορίου που τώρα συνοδεύουν τις δραστηριότητες εμπορικής πολιτικής της Ένωσης προηγούμενα ε, ήταν κατά του ΠΟΕ. Αυτές ήταν τότε, εκείνο τον καιρό, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις ήταν το μόνο φόρουμ για εμπορική πολιτική και εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις φαίνεται να αγγίζουν τις ζωές των ανθρώπων πιο άμεσα, όπου έφαίνεται πιο απομακρυσμένο, αλλά εμείς αισθανόμαστε αλληλεγγύη με όσους χρειάζεται να εξηγήσουν την εμπορική πολιτική σε ένα ε, ταραγμένο ακροατήριο. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και η εμπορική πολιτική προσπαθεί να σχηματίσει, να σχεδιάσει την παγκοσμιοποίηση έτσι ώστε να είναι υποφελή για όλους. Η προσέγγιση με βάση την αξία θα πρέπει αυτό να το καταστήσει δυνατό το εμπόριο για όλους είναι μια αξιόπιστη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρου τον κόσμο, υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη διατήρηση των δημοσίων υπηρεσιών και τον χώρο πολιτική. Είναι αλήθεια ότι το εμπόριο για όλους αυτό ε, το ορίζει πολύ ξεκάθαρα, αλλά δεν είναι νέο χαρακτηριστικό τη Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική όπω εμεί την παρατηρούμε από τον ΠΟΕ. Στον ΠΟΕ αυτή η προσέγγιση που καθοδηγείται από τι αξίε ε, καθέστη εμφανή στο ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλέ ομάδε εργασία για την προσχώρηση νέων μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε το κύρο αυτών των διαπραγματεύσεων ώστε να ορίσει του όρου εισδοχή νέων υποψηφίων με την εσωμάτωση νέων ε, προδιαγραφών. Κάποιε ε, φορέ αυτό οδήγησε σε σημαντική παράταση των διαπραγματεύσεων, αλλά πιστεύω πω ήταν αυτό προ όφελο όλων. Όταν το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαψε να είναι ο τελευταίος πιστός μαθητής του πολυμερούς συστήματος και αποκλειστικά και της πολυμερούς προσέγγισης αποκλειστικά ώστε να ξεκινήσει νέες διμερείς διαπραγματεύσεις πέρασε μια μακρά περίοδο χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα μόλις ακούσαμε πως αυτή η περίοδος φαίνεται να κλείνει πια και ε, φαίνεται ότι αποκομίζεται τα ωφέλη αυτού του μόχθου. Εγώ τολμώ να προτείνω ότι άλλες χώρες που διαπραγματεύονται, ας πούμε με τη, τα κράτη ΑΣΕΑΝ, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα γιατί ήταν λιγότερο φιλόδοξα. Λιγότερο φιλόδοξα όχι μόνο όσον αφορά την κάλυψη προϊόντων, αλλά και όσον αφορά την θέσπιση ορισμένων αξιών. Άρα λοιπόν θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι στις διαπραγματεύσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε την θυσία των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων προς χάρη μιας προσέγγισης που, θα που οδηγείται, καθοδηγείται από αξίες. Οι καλές ιδέες συνήθως προηγούνται τον καιρού, του καιρού τους. Ένα παράδειγμα είναι τα θέματα της Σιγκαπούρης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρότεινε, χρειάστηκε μετά να τα εγκαταλείψει στο Κανκούν και τώρα επανέρχονται μπορεί και επενδύσεις είναι ένα παράδειγμα. Μόνο τώρα αρχίζει ο κόσμος να εκτιμά την, το πόσο σκόπιμο είναι να αναπτυχθούν και αρχίζει να δίνει χώρο για αυτά σε πολυμερές επίπεδο. Και αυτό ίσως προκαλείται από την εμπειρία που κερδίθηκε στις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες. Η εμπορική ατζέντα λοιπόν της Ένωσης είναι ευπρόσδεκτη λοιπόν στον ΠΟΕ γιατί στρώνει το δρόμο για τις μελλοντικέ πολυμερείς προσεγγίσεις. Οι διμερείς και οι περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν τα πραγματικά, τα πραγματικά θεμέλια για τις πολυμερείς συμφωνίες. Το σημερινό πρόγραμμα, όπως ε, το βλέπουμε σήμερα, λέει Ευρωπαϊκή Ένωση ίσον ο σχεδιαστής της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω και ένα θαυμαστικό στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, thank you. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας αυτή. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ζωντανή ε, συνεδρία ερωταπαντήσεων στη συνέχεια, αλλά πριν από αυτό έχουμε ακόμα δύο σημαντικές συμβολές από τον ΠΟΕ. Να περάσουμε στο δούνο Και οι δύο θεσμοί βεβαίως συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίσουν την λειτουργία, την ορθή λειτουργία του, του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος και του συστήματος πληρωμών. Έχουμε αυτόν τον ε, διασυνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε και φυσικά ο ρόλος του Δουνουτού για το εμπόριο δεν μπορεί να παραμεληθεί. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Τζέφρι Φρανκς που είναι διευθυντής των γραφείων του Δουνουτού για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ τα μέλη του Κοινοβουλίου, την Επίτροπο, τους διακεκριμένους προσκεκριμένους που βρίσκονται εδώ. Είναι μεγάλη τιμή της πρόσκλησης που μου απευθύνατε Έχουμε προσπαθήσει και με την Κριστίν Λαγκάρτ από το Διεθνέ Ταμείο να προσεγγίσουμε μέσω του κοινοβουλευτικού δικτύου και σα έχουμε διανύμει τι σχετικέ πληροφορίες τους βουλευτέ ε, όλων των κοινοβουλίων γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμη η συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό, ε, την Υπηρεσία συγγνώμη, Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια εκδήλωση που έρχεται την, σε κρίσιμη στιγμή. Έχουμε μια μακροχρόνια συνένεση μεταξύ οικονομολόγων ότι ένα πιο ελεύθερο εμπόριο είναι θετικό για την παγκόσμια εμπόρια. Με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς προσκόμματα μπορούν και οι πόροι να χορηγηθούν, να κατανεμηθούν στην καλύτερη τους δυνατή χρήση, να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις επιλογές για τον καταναλωτή. Για πολλά χρόνια αυτή η πεποίθηση, η οικονομική πεποίθηση υποστηρίχθηκε από μια ευρεία πολιτική πολιτική συνένεση, πολιτική υποστήριξη που έκυψε ύστερα από τι καταστροφικές εμπειρίες του προστατευτισμού και τη μεγάλη ύφεση έχει οδηγήσει και στη σύσταση της Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ε, την ίδρυση των διεθνών οργανισμών όπως Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ε, Διεθνού Νοσηματικού Ταμείου. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε και εδώ στην Ευρώπη στην δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ε, ε, αλλεπάλληλους γύρου της ΓΑΤ για τις διαπραγματεύσεις στο εμπόριο. Πρόκειται για μια πολιτική συνένεση όμως για τη διαμόρφωση ενός ε, πιο ελεύθερου εμπορίου που τώρα όμως υποχωρεί. Ο γύρος της Ντόχα δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν με την, συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά ήταν μια αντιμετώπιση σημαντική αντίσταση και πολύ μεγαλύτερη αντίσταση και ε, αντιμετώπισε και η συμφωνία TTIP ε, και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. η εταιρική σχέση του ειρηνικού αντιμετώπισε σε επίπεδο των δύο σωμάτων της Αμερικανικής Βουλής πολύ μεγάλη αντίσταση και βέβαια μια σκληρή απόφαση Brexit, Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις από το ελεύθερο εμπόριο. Ταυτόχρονα βλέπουμε σημαντική ε, μείωση στο ποσοστό ανάπτυξης στο παγκόσμιο εμπόριο. Από το 2012 η ανάπτυξη ε, στο εμπόριο ε, προϊόντων και υπηρεσιών ε, έχει περιοριστεί στο 3%. Τι συμβαίνει λοιπόν ως προς την οικονομική πτυχή. Έχουμε πρόσφατες έρευνες από το Διεθνές Μασματικό Ταμείο που δείχνουν ότι τα 3 τέταρτα των ελλημάτων που σημειώνονται στο Διεθνές Εμπόριο από το 2012 μπορούν να αποδοθούν σε υποβαθμισμένες επενδύσεις μικροοικονομική δηλαδή, μικροοικονομικά προβλήματα στην ανάπτυξη. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ε, πορεία της απελευθέρωσης του εμπόριου που είναι αρκετά βραδία. Δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενίσχυση αυτών των συναλλαγών και μετά την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση αναδύονται φραγμοί στο εμπόριο που μπορούν να αποτελέσουν επιπλέον κινδύνους. Η επανεγκατάσταση μεγάλων ε, επιχειρήσεων, μεγάλων αλυσίδων παραγωγής, ε, η αναζήτηση χαμηλότερου κόστου στην παραγωγή δεν δίνουν μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα ως προς το εάν έχουν εξατληθεί αυτές οι δυνατότητες της αλυσίδας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο ή αν απλώς έχουν υποβληθεί στις πιέσεις σε σχέση έχουν παρεμποδιστεί από τις πιέσεις σε σχέση με το ελεύθερο εμπόριο. Η οικονομία λοιπόν μπορεί να αναζωογονηθεί, αλλά ανάπτυξη δεν αναμένεται να εμφανιστεί σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της περίοδου πριν από την οικονομική κρίση, εάν δεν αναπτυχθούν περισσότερο οι αλυσίδες παραγωγής αξίας. Και βέβαια σε σχέση και με την Κίνα βλέπουμε ότι περιορίζεται η δυνατότητα που είχαμε στο παρελθόν και επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Η οικονομική πτυχή ήταν αυτή, η πολιτική πτυχή τώρα, ε, με σημαντική δυσφορία που εκδηλώνεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, από εκείνου που θεωρούν ότι έχουν χάσει το παιχνίδι, τον αγώνα δρόμου του παγκόσμιου εμπορίου. Ε, ναι, δεν ε, μπορούμε να αρνηθούμε ότι παράγει απώλειες, όχι μόνο κέρδος στο παγκόσμιο εμπόριο, για εκείνου όμως οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις διάφορες χώρες που δεν είχαν επαρκή προστασία έναντι της χρήσης πιο ελεύθερων συνθήκων εμπορίου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τις πιο ανεπτυγμένες κοινωνίες ή των συνθήκων εργασίας σε άλλες. Όπως είπε και η Επίτροπος Μάλμστρομ, οι διαπραγματευτές συμφωνιών όπως ε, η ΣΕΤΑ, όπως η TTIP, η TTP έχουν ε, αποκομίσει τα διδάγματα και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια, στην προστασία των εργαζομένων, των περιβάλλων, στι νέε αυτέ συμφωνίε. Αλλά βλέπουμε ότι πολέμοι αυτών των συμφωνιών αντιδρούν χωρί καν να δουν την ουσία των αποφάσεων και των προτάσεων. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε να συνεχίζονται οι πιέσεις ως προς την οικονομική ανάπτυξη και να μην δίνεται επαρκής οικονομική απάντηση στις ε, ε, ανάγκες. Το εμπόριο μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερη ανάπτυξη και κέρδος για ολόκληρο τον κόσμο. Νέες τεχνολογίες, νέες διαδικασίες από ξένες αγορές που αποτελούν πηγή πλούτου. Υπάρχει περαιτέρω βέβαια περιθώριο για την ε, για τον περιορισμό των τελωνιακών δασμών που έχουν παραμείνει, για την διευκόλυνση περισσότερο των εμπορικών συναλλαγών για μια πορεία ε, πρόοδου για το γύρο της ντόχας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε στους τομείς που έχουν μεγαλύτερη σημασία και αξία για τις οικονομίες, υπηρεσίες, συνεργασίες, ε, διασυνοριακές επενδύσεις και εμπόριο και νέες συμφωνίες όπως τη ΣΕΤΑ. Στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό αυτοί οι στόχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό παράδειγμα και υπόδειγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια μελλοντική εμπορική συνεργασία για άλλες περιοχές του κόσμου. Οι συνολικέ συμφωνίε εμπορίου που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά, τι ΗΠΑ αλλά και άλλε ζώνε του κόσμου, όπω είπε και η Επιτροπό, μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον πλούτο για τι περιοχέ αυτέ η ολοκλήρωση αυτή η εμπορική ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στις ανησυχίες των εργαζομένων που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Θα πρέπει να διευκολύνει την προσαρμογή και τη μετάβαση με ε, ευραία δίκτυα προστασίας, με κατάρτιση, με ανάπτυξη δεξιοτήτων, με διευκόλυνση της γεωγραφικής αλλά και επαγγελματικής κινητικότητας. Αυτά τα δίκτυα ασφαλείας τα έχει κατά τον καλύτερο βαθμό επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να αποτελέσει πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο παράδειγμα για τους άλλους, για το πώς το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να αποβεί ει όλων των πολιτών και δι των Ευρωπαίων. Έχει πληγεί από την ε, οικονομική κρίση Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί Ευρωπαίοι αισθάνονται δυσφορία από την βραδία ανάκαμψη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι να γυρίσουμε την πλάτη στις πολιτικές που μπορούν και έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να καταστήσουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πλούσια το διεθνέ εμπόριο, έχει μπορέσει να βγάλει από τη φτώχεια εκατομμύρια Κινέζων, έχει δώσει νέους πόρου σε εκατομμύρια πολιτών στην ε, Λατινική Αμερική και πρόσφατα και την Αφρική. Και όπως ε, αναφέρθηκε ο Μπομπ Ντίλαν από τον κύριο Βίνκλερ, θα συνεχίσω και εγώ στην ίδια, ε, στον ίδιο ρυθμό. Ναι, αλλάζουν οι καιροί, λέει ο Μπομπ και συνεχίζει. Εάν ανεβαίνουν τα νερά, και βρέχεσαι μέχρι το κόκαλο, ήρθε η ώρα να κολυμπήσεις, αλλιώς θα βυθιστείς σαν την πέτρα. Ναι, αλλάζουν οι καιροί. Και όσο ε, ανεβαίνουν τα νερά, πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε, πρέπει να αρχίσουμε να κολυμπάμε. Και όπως είπε η Διευθύντρια του Διεθνούς Οικονομικού Ταμείου, κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, πρόσφατα, μπορεί τώρα να βλέπουμε μεγάλη αντίθεση, αλλά ακριβώς τώρα είναι η στιγμή που χρειάζεται περισσότερη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που χρειάζεται ο κόσμος. Περισσότερη συνεργασία λοιπόν και όχι λιγότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φρανξ για την συμβολή σας στην συζήτηση και για αυτό το όραμα για το μέλλον που είμαι βέβαιος ότι πολλοί συμμερίζονται. Θα ακολουθήσει ένας από τους πολύ σημαντικούς εταίρους του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η, η Επίτροπος μίλησε για τον φάκελο των ορυκτών που προκαλούν συγκρούσεις. Και ε, υπάρχει μελέτη του ΩΣΑ και γι' αυτό χαίρομαι που είναι κοντά μας ο κύριος Κεν Άσ. Έχει τον λόγο από τον ΩΣΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και εσείς κυρία Επίτροπε και ε, εσείς οι άλλοι συνάδελφοι επιθυμώ να πω λίγα λόγια που δεν αφορούν μοναχά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πάντως ε, την αφορούν και να εξηγήσω ιδίω γιατί πιστεύουμε ότι το εμπόριο περνάει δύσκολους καιρού σήμερα. Θα πω και λίγα λόγια σχετικά με το τι ίσως θα θέλαμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Στο οικονομικό επιχείρημα νομίζω ότι ο Τζέφρι Φράνξ εξήγησε το έργο που κάνουν οι συναδελφοί μας και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, υπάρχει ένα γεγονός όμως. Περνούμε τώρα την ε, μεγαλύτερη περίοδο στασιμότητας στο ε, παγκόσμιο εμπόριο από τη δεκαετία του 70. Πρόκειται για μια φάση η οποία είναι μοναδική και σε ό,τι αφορά το βάθος και τη διάρκεια. Κάτι που ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι το εμπόριο αντιμετωπίζει ε, αντίθετους άνεμους, κυρίως τις επιφυλάξεις του κοινού και αυτό που έδειξε και η πρόσφατη αμερικανική εκλογή είναι μια αντίδραση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού που θεωρούν ότι βλάπτονται από ε, την πρόθεση του διεθνούς εμπορίου αντί να κερδίζουν. Όμως, όπως εξήγησαν και άλλοι προηγουμένως, το εμπόριο έχει προωθήσει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόληση όλες τις οικονομίες μας. Και το εμπόριο εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινή ζωή μας από τα τρόφιμα που έχουμε στο τραπέζι μας, τα φάρμακα που μας κρατούν υγιείς, τα διάφορα ευφυή, τηλέφωνα και όλα αυτά που εσείς παίζετε, ορισμένοι από εσάς που εξακολουθούν και παίζουν την τελευταία ώρα, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε το εμπόριο. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να συμφιλειωθεί αυτή η κατανοητή ίσως επιφύλαξη του κοινού και η οικονομική συνένεση που περιγράφεται από την άλλη μεριά. Ας είμαστε ειλικρινεί. Με κάποιους τρόπους έχουν δίκιο αυτοί που είναι επιφυλακτικοί. Τα πλεονεκτήματα του εμπορίου δεν ωφελούν τους πάντες και πάντοτε. Και ούτε τα ε, ωφελήματα είναι άμεσα ορατά. Υπάρχουν και άνθρωποι ή και περιοχές που πλήττονται ε, κυρίω εκείνοι οι οποίοι έχουν την μικρότερη ικανότητα για να προσαρμοστούν. Όμως, από άλλη άποψη, αυτοί που είναι οι σκεπτικιστές δηλαδή ε, είναι, έχουν απόλυτος άδικο. Δηλαδή, η απομόνωση σημαίνει απομόνωση και της κοινωνίας από νέα προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες. Τα προστατευτικά μέτρα δεν προστατεύουν στην πραγματικότητα ούτε τα άτομα, ούτε τις εταιρείες, ούτε τις περιφέρειες. Αντίθετα, τα φορτώνουν κόστος και εμποδίζουν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε νέα ανάπτυξη και σε νέα προϊόντα. Με πολλούς τρόπους η οικονομική συνένεση επίσης έχει κάποιο δίκαιο. Δηλαδή, οι ανοιχτές οικονομίες όντως αναπτύσσονται ταχύτερα από κλειστές οικονομίες. Μισθοί και συνθήκες εργασίας είναι πάντοτε καλύτερες, σχεδόν πάντοτε καλύτερες σε εταιρείες οι οποίες διεξάγουν εμπόριο από ό,τι σε αυτές που δεν διεξάγουν εμπόριο. Μέσα από τις δεκαετίες το εμπόριο πήρε από το χέρι εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων και τους έβγαλε από την φτώχεια. Όμως επίσης είναι λάθος να ισχυρίζεται κανείς ότι η εμπορική πολιτική και από μόνη της θα ωφελήσει όλο τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει η απασχόληση, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και οι άνθρωποι, οι οικογένειες που έχουν μικρό στενό προϋπολογισμό. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι το εμπόριο θα ωφελήσει όλους μόνο εφόσον οι κυβερνήσεις υιοθετήσουν και τις διαρθρωτικές εκείνες πολιτικές που θα επιτρέψουν στις οικονομίες να λειτουργήσουν αποδοτικά και οικονομικά. Από τη λειτουργία των αγορών μέχρι τις στατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις φυσικές, στις, ε, φυσικές υποδομές και ούτω καθεξής. Δηλαδή η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κενό. Θα πρέπει να αποτελεί, αποτελέσει τμήμα του ιστού των ε, εγχωρίων πολιτικών. Μπορούν λοιπόν οι κυβερνήσει να κάνουν πολλά πράγματα. Πάλι ο Τζέφρι είπε σχετικά με τα ε, όργανα που είναι δυνατόν να, να χρησιμοποιηθούν. Η νομισματική πολιτική δεν υπάρχει πολλή χώρος πλέον εκεί. Στα δημοσιονομικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημοσιονομική πολιτική για να ενισχύσει την ανάπτυξη και τα ωφελήματα από αυτήν. Όμω οι κυβερνήσει μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα. Δύο θέλω να πω πιο συγκεκριμένα. Και εδώ δεν μπορείτε να επιλέξετε πρέπει να κάνετε και τα δυο. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, και πάλι αυτό λέχθηκε προηγουμένως, πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην μείωση των περιττών εξόδων, του περιττού κόστους στο εμπόριο. Και μπορούν να το κάνουν αυτό αποφεύγοντας να λάβουν νέα προστατευτικά μέτρα ή κάνοντας απλά πράγματα. Βελτιώνοντας, για παράδειγμα, τις μη αποδοτικές τελωνιακές διαδικασίες που υπάρχουν ακόμη ανάμεσα στα σύνορά μας. Να αντιμετωπίσουν ή να μειώσουν τους δασμούς σε ορισμένους τομείς και άλλα μέτρα, για παράδειγμα, που διέπουν πολλές, πολλούς τομείς υπηρεσιών. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις της εγχώρηση στις ε, εσωτερικές πολιτικές τους για να υποστηρίξουν ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που υπάρχουν στις διάφορες χώρες, στις επιμέρους χώρες. Τα συστατικά είναι γνωστά. Η συνταγή θα είναι διαφορετική αναχώρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις έμφαση πρέπει να δοθεί στην βελτίωση της ικανότητας των εργαζόμενων και των αγορών να αντιμετωπίσουν, να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, υποδομές κτλ. Από την άλλη μεριά, σε άλλες περιπτώσεις η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε ενίσχυση των κοινωνικών δομών για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και οικογένειες που δεν είναι τόσο εύκολο να προσαρμοστούν. Αυτά είναι δύο σκέλη των ίδιων στόχων. Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να ληφθούν στο εθνικό επίπεδο. Οι κυβερνήσει όμω μπορούν να καταβάλουν προσπάθειε και να διαπραγματευτούν και το πράττουν άλλωστε αυτό και νομικά δεσμευτικέ, περιφερειακέ, πλειονομερεί αλλά και ιδίω πολυμερεί εμπορικέ συμφωνίε για να θεμελιώσουν αυτές τις εθνικές στρατηγικές. Όχι επειδή μας αρέσει να θεμελιώνουμε ή να κρίνουμε πράγματα, αλλά διότι θέλουμε να υπάρχει προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές. Αλλά ταυτόχρονα και για να επεκταθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, διανέμοντας έτσι τα ωφέλη σε περισσότερους. Εμπορικές συμφωνίες λοιπόν μπορούν να απαντήσουν στις ανησυχίες του κοινού για την κατανομή των ωφελημάτων του εμπορίου με την αντιμετώπιση αυτών των συμπληρωματικών μη εμπορικών πολιτικών που ωστόσο έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα. Αντί λοιπόν, και ολοκληρώνω με αυτά, αντί να προσπαθούμε να ανακόψουμε την πορεία του εμπορίου, σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να προωθήσουμε ένα πιο προοδευτικό, πιο ανοιχτό, πιο συνεκτικό πακέτο επενδυτικών και εγχώριων ε, πολιτικών πιο ανοιχτών που να προσφέρουν περισσότερη απασχόληση σε περισσότερους ανθρώπους. Ο καλύτερος τρόπος θα είναι πολυμερός μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επίσης με πλειονομερείς ή περιφερειακές συνεργασίες έχουμε δει και κάποιες επιτυχίες όπως η περίφημη συμφωνία με τον Καναδά που ακούστηκε ήδη μερικές φορές. Αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Η ανικανότητα να προχωρήσεις με την ταχύτητα που ε, χρειάζεται στο διεθνές επίπεδο δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην προχωρήσεις και σε εθνικές πολιτικές. Ευχαριστώ, θα αρκεστώ σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ήταν η ώρα να στραφούμε στους βουλευτές της Επιτροπής μας για ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Καταρχάς θα δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές ως ήθιστε και για να έχουμε χρόνο για να ακούσουμε και τις απαντήσεις των διακεκριμένων μας ομιλητών θα προτείνω καθένας να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων. Συνάδελφος Φιέλνερ από το ΕΛΚΑ πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντική συζήτηση που κάνουμε σε δύσκολους καιρούς καθώς πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση γιατί βλέπουμε σήμερα το θέμα του εθνικισμού και του προστατευτισμού. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τον Τραμπ, αλλά σαφώς είναι της μόδας ολόκληρο τον κόσμο του ίδιου είδους εθνιστικές και λαϊκιστικές ηγεσίες. Και εμείς εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα αγωνιστούμε θα, κατά αυτών των ιδεών ή θα προσπαθούμε να ε, ε, αντιδράσουμε διαδίδοντας τις ορθές ιδέες. Έχω την αίσθηση ότι η παγκοσμιοποίηση κατηγορείται για τα πάντα. Γι' αυτό έχω μια ερώτηση. Από τη δική μου προπτική εγώ διερωτώ με πολλές ε, από τις επιπτώσεις της ε, κατανομής του πλούτου Μήπως θα έπρεπε να μας απασχολήσει περισσότερο η νομισματική πολιτική που ε, έχουμε εφαρμόσει τελευταία και την επιπτώσεις αυτής. Δεν, δεν είναι κάτι για το οποίο ψηφίζει ο κόσμος, για την εμπορική πολιτική ψηφίζει. Εμείς ως πολιτικοί όμως δεν θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο την νομισματική πολιτική και τις επιπτώσεις αυτής. Δεύτερον, ευχαριστώ που ακούσαμε για τα όσα ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της εμπορικής πολιτικής και για τα όσα μας είπατε για τις ε, εμπορικές μας συμφωνίες κτλ. Όμως, μήπως τώρα έχουμε πάει πολύ μπροστά και αφήνουμε πίσω τις καλές ιδέες που είχαμε κάποτε. Μήπως αυτές οι συμφωνίες πια είναι τόσο βαθιές και τόσο καθολικές που δεν μπορούμε καν να τις συλλάβουμε. Η συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, ας πούμε, είναι εξαιρετικά περίπλοκη και στη βάλουμε στην άκρη. Ποιε θα ήταν οι συνέπειε για την παγκόσμια ατζέντα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποκλιμακώσει αυτές τις συμφωνίες και έπειτα αν Παγκοσμίως βλέπουμε ότι η απόλυτη φτώχεια έχει μειωθεί σε, δραματικό, σε τεράστιο βαθμό. Έχουμε ε, τέτοιου είδου τάσει και αλλού σε άλλε φτωχέ χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο David Μάρτιν από του Σοσιαλιστέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ε, ξέρουμε, η, ε, η ρητορική κατά του εμπορίου είναι και κατά τη παγκοσμιοποίηση και αυτοί που επικρίνουν την παγκοσμιοποίηση την επικρίνουν γιατί βλέπουν ότι οι φόροι ας πούμε ξεφεύγουν από το κρατικό έλεγχο αλλά δεν αντικαθίσταται ο έλεγχο αυτός από κάποιον άλλον βλέπουν ότι η διαφθορά είναι ευκολότερη διασυνοριακά Εσεί βλέπετε ότι θα, υπήρχε, θα ήταν σκόπεμο στις εμπορικέ μα συμφωνίε να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτά τα θέματα ή να μείνουμε αποκλειστικά στα εμπορικά Δεύτερο, δεύτερη ερώτηση νομίζω ο κ. Μπέρνερ το είπε αυτό, ότι συχνά πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στο μάκρο των διαπραγματεύσεων και την ποιότητα της συμφωνίας. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά διρωτώ με μήπως ε, το παρακάνουμε όταν 5,5 χρόνια περνάνε πριν φτάσουμε σε εμπορική συμφωνία. Αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο πραγματικά ή με τις διαδικασίες μήπως που είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό να δίνω και μια ερώτηση στην Σεσίλια. Πιστεύετε ότι το ΣΕΤΑ έχει υποβαθμίσει την εμπιστοσύνη σε μας ε, ως αξιόπιστο εταίρο. Ε, μήπως δηλαδή κάποιοι που θα ήθελαν να συμφωνήσουν μαζί μας ε, το ξανασκεφτούν λόγω αυτής της περιπέτειας. Τελευταία μου ερώτηση. Φιλιππίνες. Μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε τις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις εκεί γιατί περιγράφουμε τον εαυτούς μας ως μια ήπειρο που κάνει τις συμφωνίες της με τη βάση αξιών. Μήπως πρέπει να πούμε στις Φιλιππίνες ότι δεν μπορούμε πλέον να διαπραγματευτούμε και επειδή κανεί και άλλοι αναφέρουν τον Τραμπ. Αν ο Τραμπ προχωρήσει με το 25% δασμούς προς την Κίνα, που θα πούμε, ας πούμε ότι το κάνει, δεν νομίζω ότι το κάνει. Ε, μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τα αγαθά που δεν θα παίρνει πια η Αμερική και θα πρέπει να τα γεωτεκινήσουμε αλλού. Ευχαριστώ κύριο Στάρμπατη. Mm. Ως οικονομολόγος ξαφνιάζομαι δεδομένου ότι είναι βέβαιο ότι διευκολύνει το διεθνές εμπόριο την ανάπτυξη οικονομίας. Ωστόσο έχουμε μια διαφορετική εμπειρία τώρα, μια αναμφισβήτητη ε, ε, θεωρία, ένα αξίωμα, βλέπουμε τώρα να αμφισβήτηται μέσα από την πολιτική και πρέπει να δούμε σε τι οφείλεται αυτό. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προχώρησαν μεν τα πλεονεκτήματα του διεθνούς εμπορίου, χωρίς όμως αυτά, ταυτόχρονα έχει εξηγηθεί ότι συνεπαγόνται και κάποιες δυσκολίες, γιατί το άνοιγμα των αγορών σημαίνει περισσότερο ανταγωνισμό, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός σημαίνει πιο σκληρό ανταγωνισμό, περισσότερες δυνατότητες αλλά και περισσότερες χρεοκοπίες. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να πιστεύει κανείς ότι αυτόματα κερδίζουν όλοι. Θα κερδίσουν μόνοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν μια πολιτική προσαρμοσμένη στο ελεύθερο εμπόριο, με την ανάπτυξη του κεφαλαίου, με την κατάρτιση, με τη φορολογική πολιτική, με την νομισματική της πολιτική. Όλα αυτά μαζί είναι παράγοντες οι οποίοι ε, φέρνουν τελικά την, ε, το πλεονέκτημα από το, εμπο, από το διεθνές εμπόριο και νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε τονίσει, το λέω και ως οικονομολόγος αρκετά, με τη συζήτηση για τη ΣΕΤΑ που έγινε στο Στρασβούργο. Ο κύριος Λάμπερτς, συμπρόεδρος των Πρασίνων, είπε ότι το όχι της Βαλονίας ήταν ένα νέο ναι στην Ευρώπη. Για <laughs> φανταστείτε το αυτό. Μια μικρή επαρχία να μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την Ευρώπη. Η κυρία Λεπένα, η οποία λέει ότι ε, ε, μπορεί ε, με βάση κάποια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Τάφτς να βγει τελικά αποτέλεσμα αυτή η συμφωνία της ενίσχυσης ανεργίας. Μα κανείς δεν είπε ότι υπάρχουν μόνο θετικά, θετικές εξελίξεις και πλεονεκτήματα, θα υπάρξουν και μειονεκτήματα, αλλά αυτό δεν εξηγήθηκε αρκετά. Και γι' αυτό θα πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει βάση διαφοροποίησης μεταξύ της επιχειρηματολογίας των Πρασίνων και της Μαρίν Λεπέν. Είναι ακριβώς η ίδια γραμμή της επιχειρηματολογίας. Ναι, μου επιτρέπετε πρόεδρε, τελειώνω. Είναι όμως ε, οφθαλμοφανέστατο αυτό και ήθελα να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much ε, for the liberals, ε, coordinator Σας ευχαριστώ πολύ, φιλελεύθερη κυρία Σάκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ όντως έρχεται την κατάλληλη στιγμή η συζήτηση και αν λάβουμε υπόψη το ζωφερό σύννεφο που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Είναι ένα πολύ ευρύ ζήτημα αυτό του Διεθνού εμπορίου. Δεν ε, έχω την ε, ψευδέστηση ότι μπορούμε να θέσουμε ε, φραγμού στην παγκοσμιοποίηση. Όχι βέβαια. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα τη διαμορφώσουμε, τι ευθύνε μπορούμε να αναλάβουμε ώστε να την πλαισιώσουμε μέσα σε ένα σύνολο κανόνων ρεαλιστικό, σε ένα σύνολο κανόνων που θα φέρει θετικέ εξελίξει για του πολίτε. και Πρέπει να σημειώσω ότι πολύ συχνά φαίνεται ε, στο δημόσιο διάλογο να διωγγώνεται και η ελπίδα και ο φόβος του τι μπορεί να φέρει ή τι δεν μπορεί να φέρει το διεθνέ εμπόριο και ποιο είναι υπεύθυνο για την όποια εξέλιξη και αλλαγή. Πρέπει να εξυγχρονιστούν οι κανόνε για το εμπόριο, πρέπει να προσφέρουν υπηρεσία στον πολίτη, όπως άλλωστε είναι καθήκον δικό μας, και πρέπει να διαφοροποιηθούμε από αυτούς οι οποίοι απλώς θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να προβούν σε συμβασμούς και εκείνους που θέλουν να είναι κομμάτι των διαπραγματεύσεων μόνο και μόνο για να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν και στον καθρέφτη. Πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμεί. Το λέω αυτό ρητά στην Επιτροπή που βρισκόμαστε, στο Κοινοβούλιο που βρισκόμαστε, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη βεβαίω και οι εθνικέ κυβερνήσει όπω και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ευθύνη, αλλά και εμεί πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να πράξουμε έτσι ώστε να μην αποστέλουμε ε, ουτοπιστικά μηνύματα, να μην υποδαβλίζουμε μια φωτιά την οποία θα μπορέσουμε να σβήσουμε, εάν αυτή δεν ήταν τουλάχιστον η πρόθεσή μας. Και πρέπει να αντιληφθούμε τι διακυβεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή είναι η ερώτησή μου προς τους ομιλητές, των οποίων ε, κρίνω πολύ αξιόλογες τις τοποθετήσεις. Εάν το εμπόριο δεν είναι πλέον ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια δεν θα μου περνούσε καν από το μυαλό ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο και τόσο κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο. Οι ομιλητές λοιπόν τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε, ποια πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι η συγκριτική ε, ανταγωνιστική δυνατότητα και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα μπορούσε να κάνει εάν ε, δεν ήταν σε θέση να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση νέες εμπορικές συμφωνίες ανταγωνιστικά, ποια θα ήταν η θέση τη και ποια θα ήταν και οι συνέπειε, ποιε θα ήταν οι συνέπειε για την εσωτερική αγορά, αν το κάθε κράτο μέλο χωριστά ξεκινούσε τι διαπραγματεύσει για τι εμπορικέ συμφωνίε. Αυτή είναι μια ερώτηση και θα προσθέσω άλλη μία θα έχουμε δυνατότητα να διαπραγματευτούμε άλλες συμφωνίες, δηλαδή να ε, βάλουμε στην πλάστικα το ειδικό μας ε, πολιτικό και εμπορικό βάρος για άλλες συμφωνίες, για την κοινωνία της πληροφορίας, για το περιβάλλον, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε και ε, καλλιεργούμε στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πράγματι είναι επίκαιρη συζήτηση Ευχαριστώ πολύ και για τις εισρωές σας έως τώρα. Αλλά νομίζω οι ερωτήσεις, οι ερωτήσεις πρέπει να μπουν και πιο βαθιά. Παγκοσμιοποίηση και εμπόριο είναι άραγε το ίδιο. Όταν λέμε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια εμπορική πολιτική έτσι ώστε να μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι η παγκοσμιοποίηση είναι αντικειμενική διαδικασία και εκεί λειτουργούν άλλες δυνάμεις. Πώς δρούμε και πώς αντιδρούμε εμείς απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που βάζουν και τους όρους για την κοινωνική ανάπτυξη, για την ε, παραγωγή, για την κατανάλωση και ούτω καθεξής και τι, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον καθέναν από εμά. Αυτή νομίζω είναι μια πρόκληση που πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν θέλω ωστόσο να αποκλίνω από τα βασικά, γι' αυτό θα κάνω δύο ερωτήσεις. Ανάπτυξη που αναφέρθηκε πριν για τους περισσότερους ανθρώπους δεν σημαίνει ωστόσο αύξηση της προσωπικής τους ευημερίας είπατε και πριν, ότι υπάρχουν και πολλοί χαμένοι από την εφαρμογή της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Βλέπουμε επιταχυνόμενη σόρευση κεφαλαίου μεταξύ των πλουσίων και επιδίνωση άλλων παραμέτρων. Και η εναλλακτική επιλογή για μένα είναι το fair trade, το έντιμο δίκαιο εμπόριο. Δηλαδή επιστροφή σε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους φτωχότερους παραγωγούς. Η αρχιτεκτονική που ακολουθείται τώρα δεν αφήνει χώρο για το έντιμο δίκαιο εμπόριο και κυρίως σε ό,τι αφορά την, τον προσανατολισμό των διαδικασιών προς εκεί όπου είναι δυνατόν να υπάρξει το fair trade και σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες παραγωγής στις ε, χώρες όπου μπορούν να ενδιαφέρονται. Άρα, τελικώς η κανονικότητα είναι το unfair trade και γι' αυτό πώς θα το αλλάξουμε. Δεύτερο, η δημοκρατική διάσταση. Δεν φτάνει να δηλώνουμε δεν φτάνει να, μάλλον να, να εξηγούμε εμεί του ανθρώπου, εμεί εδώ οι ευρωβουλευτέ εκπροσωπούμε και τα συμφέροντα των ψηφοφόρων. Άρα πρέπει να περιλάβουμε, πρέπει να μεταφέρουμε εδώ τι απόψει του για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Βίνκλερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν πράγματι καλή ιδέα να σεβαστείτε όλοι τα δύο λεπτά, διότι αναμένουμε βέβαια με μεγάλη ανυπομονησία τις απαντήσεις των ε, αξιότιμων μελών, των διακεκριμένων μελών του πάνελ. Ο κ. Μπούχερ των Πρασίνων. Έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Άρθρο 207 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού το καθορίζει. Όμως, καθορίζει ότι συνάπτονται εμπορικές συμβάσεις. Οι νέε σε βάθος συμφωνίε είναι κάτι διαφορετικό, διότι μπαίνουν βαθιά στις δημοκρατικές δομές των χωρών μελών και στα δικαιικά του συστήματα. Υπενθυμίζω την ΣΕΤΑ ως παράδειγμα και εκεί το κεφάλαιο περιρυθμιστική συνεργασίας. Εδώ οι αποφάσεις για την ομοθεσία των χωρών μελών περιορίζονται με μια λέξη, δηλαδή το «ανέστασε», το περιτό. Μπορεί κανεί να διαφωνήσει σχετικά με την ερμηνεία, αν δηλαδή θα ερμηνευτεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Αμερικανικού δικαίου, που είναι απολύτω διαφορετικό βεβαίω από το Γερμανικό δίκαιο. Ανεξαρτήτω τούτου, ό,τι και να αποφασιστεί, το ζήτημα είναι ότι την ερμηνεία θα δώσουν τα διαιτητικά δικαστήρια. Και τα διαιτητικά δικαστήρια είναι γνωστό πώ το πράττουν. Μεταρρυθμίσατε τα διαιτητικά δικαστήρια στο International Court System σαφής βελτίωση. Όμως πρέπει να, είμαστε, πρέπει να έχουμε σαφώς υπόψη ότι αυτό το court system δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που θέτουν οι διάφορες συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δικαστήριο ή σε δικαιοδοσία. Άρα, εδώ υπάρχει ακόμα χώρος για πάρα πολλές βελτιώσεις. Τονίζω και πάλι ότι οι νέες αυτές συμφωνίες τροποποιούν τη δημοκρατική και δικαιική δομή των χωρών μελών. Αυτό πρέπει να αλλάξει, εάν θέλουμε να αποφύγουμε τις μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων. Ευχαριστώ. Έξι ακόμη εγγεγραμμένοι ομιλητές. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο των εγγεγραμμένων. Ο ε, συνάδελφός μας Προύστ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτού τη ε, συνεδρίαση που είναι εντελώ επίκαιρη δεδομένη τη επικαιρότητα. Ελεύθερε συναλλαγέ, απελευθέρωση, παγκοσμιοποίηση. Αυτοί οι όροι έχουν ε, ε, πολύ έννοια και θα έλεγα ότι για μας είναι σημαντικό να ρυθμίσουμε αλλά και να αναζητήσουμε κομμάτια της αγοράς εκτός. Όπως είπατε, το ποσοστό ανάπτυξης είναι 0 με 2 στην Ευρώπη και αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να την αναζητήσουμε στις χώρες ε, της ανάπτυξης με την προϋπόθεση βέβαια της διαπραγμάτευσης σωστών ε, συμφωνιών και συγχαίρω την κυρία Μάλστρομ για τη διαπραγμάτευση με τη ΣΕΤΑ γιατί και ορίσαμε κόκκινες γραμμές οι οποίες στηρίθηκαν και πάμε προς συμφωνίες ε, όπου όλοι είναι κερδισμένοι. Ε, ε, όμως οι ελεύθερες συναλλαγές, εδώ διαφωνώ μαζί σας με αυτή τη νέα μορφή συμφωνίας, ε, δεν έχουμε άγριο φιλελευθερισμό. Πρόκειται για συμφωνίες που στόχο έχουν ακριβώς να ρυθμίσουν αυτές τις συναλλαγές, να μας προστατεύσουν και αυτό είναι και ο στόχος. Ναι, να βρούμε ναι, κομμάτια της αγοράς, αλλά με αμοιβαιότητα, με κανόνες για να δημιουργηθεί ένα ε, κατάλληλο έφορο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις μας που επιτρέπουν τη διείσδυσή τους σε αυτές τις αγοράς. Αλλά πρέπει να καθησυχάσουμε τον πληθυσμό, να καθησυχάσουμε τα κοινοβούλια γιατί δυστυχώς χάνουμε στο σύνολο αυτών των θεμάτων για την, τον αγώνα της επικοινωνίας. Γιατί συχνά είμαστε στο, στο σημείο της καρικατούρας ε, και της παραπλάνησης. Ε, βέβαια, να θέσω τρεις ερωτήσεις και βέβαια έχουμε και τον Τόναλτ Τραμπ που έχει μια γλώσσα που συχνά βλέπουμε βέβαια τους πολιτικούς ε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη όσα λένε προεκλογικά και την πραγματικότητα μετά. Λέει ότι θέλει να φύγει από τον ΠΟΕ, ότι θέλει να κάνει φραγμού προστατευτισμού. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μέλλον τη TTIP. Ε, δεύτερον, στο βαθμό που τώρα πρέπει συστηματικά να διαβουλευόμαστε με τα εθνικά κοινοβούλια, είναι σημαντικό, αλλά θα έπρεπε ίσω να ξαναδούμε του κανόνε που συνδέονται με την ομοφωνία. Και τρίτον, αναφέρατε κάποια μέτρα για την Κίνα περιμένουμε λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα είναι ένα σημαντικό ε, θέμα δεδομένου του χρονοδιαγράμματος, ιδιαίτερα με την αντιστροφή της υποχρέωσης ε, απόδειξης. Ευχαριστώ Ποκού. Η κυρία Ροντρίγκε, ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης και για την ποιότητα όλων των παρεμβάσεων. Πιστεύω πως η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση ε, ε, δεν ε, δημιουργεί και η απάντηση μάλλον στην παγκοσμιοποίηση δεν είναι ο προστατευτισμός. Είναι όμως σημαντικό να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέσο που θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που αισθάνονται οι συμπολίτε μας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Μπορούμε να απαντήσουμε στις θεμετές ανησυχίες και τις λογικές ανησυχίες των συμπολιτών μας αν μπορέσουμε να συντονίσουμε τη διεθνή πολιτική με την εθνική πριν αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Μπράουνερ, δεν μπορούμε να ε, ρίχνουμε στην εμπορική πολιτική ευθύνες για τα όσα δεν είναι υπεύθυνοι. Όμως οι πολίτες, ε, ε, αυτό που προσάπτουν στους πολιτικούς και στους σεισμούς είναι ότι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Και ο τρόπος με τον οποίο και αυτό θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας είναι πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το συντονισμό λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις ε, αρμοδιότητες του καθενός. Για παράδειγμα, στο θέμα της μεγαλύτερης ε, μπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων και αυτά που είπε η Επίτροπος ε, είναι πολύ σημαντικά και των κρατών Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να μαθαίνουμε την εντολή για μια διαπραγμάτευση μέχρι ότου να αποφασίσει το Συμβούλιο με ομοφωνία. Δεν είναι δυνατόν τα εθνικά κοινοβούλια να μην έχουν υπόψη τους καν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν ενημερωθεί, να έχουν εμπλακεί, να είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται, υποχρεωτικό να ενημερώνονται για την πορεία των διαπραγματεύσεων και να κάνουν και έναν απολογισμό και εκπρόσωποι των εθνικών, των ευρωπαϊκών θεσμών να παρουσιάζονται και ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα φτιάχνουμε θέσεις απασχόλησης, ότι ο, ότι ο κόσμος θα μπορέσει να έχει καλύτερες δυνατότητες, καλύτερη, καλύτερους όρους διαβίωσης. Θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να προωθούμε και τις άλλες πολιτικές που θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς. Ευχαριστώ. Ο Σον Κέλλη τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την πολύ σημαντική συζήτηση ιδιαίτερα τη σήμερον ημέρα. Να, να συγχαρώ την Επίτροπο Μάλστρομ καταρχάς γιατί πέρασε τη ΣΥΤΑ μετά από 7 μακρά χρόνια διαπραγματεύσεων. Εδώ πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα και θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Δεδομένου ότι οι διαπραγματευτές εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν δηλαδή, με την εντολή των κρατών μελών και τα κρατημέλη και, το, και, το, και τα κρατημέλη που διαπραγματεύονται, βασικά στόχος τους είναι να κάνουν καλή δουλειά για τους πολίτες, να αυξηθεί το εμπόριο για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πώς γίνεται αυτή η δέσμευση ιδιαίτερα σε σχέση με τη ΣΕΤΑ και το TTIP, τώρα παρουσιάζεται ως κάτι που είναι τελικά κατά του λαού, κατά του μέλλοντος και των μελλοντικών προοπτικών των πολιτών. Και πώς ε, μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την ερμηνεία και όταν αρχίζουμε να τη διαπραγμάτευση για μια εμπορική συμφωνία να περνάμε το μήνυμα ότι είναι για το εμπόριο προς όφελος όλων των χωρών μας και όλων των, συμπολιτών μας. Είναι σημαντικό ότι χάσαμε αυτό το επιχείρημα και πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Δεύτερον, δεδομένων των διαφόρων δηλώσεων του κυρίου Τραμπ για το εμπόριο τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε σε σχέση με το TTIP. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Μοντέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώ πηγαίνετε γίνεται σήμερα η συζήτηση, γιατί όλοι αισθανόμαστε μια κάποια κατάθλιψη ύστερα από τι εκλογέ στι ΗΠΑ. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ελεύθερη συναλλαγή ήταν στο επίκεντρο αυτή τη προεκλογική εκστρατεία στι ΗΠΑ. Και αυτό διότι οι Αμερικανοί ξέρουν τι έφεραν, ε, τι συνέπειε έφεραν οι, ε, οι συμφωνίες που είχαν γίνει με κακή διαπραγμάτευση. Αυτές οι παραδείγματι ε, τη συμφωνία με το Μεξικό και τον Καναδά τη ναύτα έφεραν καταστροφικέ συνέπειε για όλου. Βεβαίω, είπατε, θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από μια συμφωνία. Ναι, αλλά είναι πολύ, λιγότεροι, είναι πολύ περισσότεροι χαμένοι από του κερδισμένου και μάλιστα οι κερδισμένοι είναι πάντα οι ίδιοι. Η κυρία Μάλμστρομ έχει προσπαθήσει κάπω ε, να επιφέρει μια αναλλαγή, αλλά και του το έχουμε επισημάνει, οι διαπραγματεύσει γίνονταν για χρόνια χωρί καμία διαφάνεια, σαν να είχαμε κάτι να κρύψουμε. Σαν να είχατε κάτι να κρύψετε και τελικά ο κόσμο πιστεύει ότι πράγματι κάτι υπάρχει που πρέπει να αποκρυφτεί. Λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματικέ συναλλαγέ, πρέπει να περάσουμε μέσα από μια επανάσταση τη διαφάνεια που θα ξεπεράσει αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν λέω ότι η κυρία Μάλστρομ είναι ε, ε, δρά εν κρυπτό όπως ο κύριος Δεγκούχ το προκάτοχό τη. Όχι βέβαια, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να επιτρέψει τη συνεργασία όχι μόνο των πραγματευτών και τεχνοκρατών αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του απλού πολίτη, των βουλευτών. Αυτό που διερωτάτε τι συμβαίνει, εν πάση δεύτερον και τρίτον, τέταρτον. Βλέπετε υπάρχουν λόγια ανησυχία και τελευταίο, εν Υπάρχει και ένας δογματισμός ε, της θεωρίας του, ε, των ελεύθερων συναλλαγών. Μιλώντας με φιλελεύθερους ε, συναδέλφους πολλές φορές, βλέπω να θεωρούν ότι είναι αυτονόητα θετικό πράγμα οι ελεύθερες συναλλαγές. Ε, όχι. Μια συμφωνία είναι καλή ή όχι. Ανάλογα με το πώς έχει γίνει η διαπραγματευσή της. Αυτό πρέπει πάντοτε να αξιολογείται. Μερικέ φορέ όντω χρειάζεται προστασία, Χωρί να θεωρείται εθνικισμό αυτό, ούτε προστατευτισμό. Χρειάζεται προστασία. Για να κοιτάξουμε τα, τη συζήτηση για τα μέσα εμπορική προστασία. Με καταθλίβει το γεγονό ότι υπάρχουν ε, κυβερνήσει στο Συμβούλιο που δεν θέλουν να προστατευτεί η Ευρώπη εναντί του, διεθνών, του διεθνούς ανταγωνισμού, να είναι ο, ο, ο, του χωριού δηλαδή η Ευρώπη στο παγκόσμιο αυτό χωριό. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, κύριος Πάμπριξ. Ε, ναι, όντως ε, είναι πολύ εύθετος ο χρόνος συζήτηση αυτής της εμπορικής πολιτικής ε, την ημέρα που ακολουθεί τις εκλογές της ΗΠΑ που οδήγησαν σε αποτελέσματα τα οποία μας κατέπληξαν οπωσδήποτε όλους και ορισμένους, ε, μπορεί, για ορισμένους μπορεί να ήταν και μια σημαντική νίκη. Εν πάση περιπτώσει, θα θέλατε να μου κάνετε κάποια σχόλια οι ομιλητές για το πώς θα βλέπατε να πρέπει να διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να επιτύχει. Γιατί πιστεύω πάντα, έστω και αν είμαι μειονοψηφία εδώ, γι' αυτό σας ζητώ να σχολιάσετε, ότι η απόφαση πολιτική, όχι νομική, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δηλώσει πως ήταν μεικτή συμφωνία, η ΣΕΤΑ, ήταν πολιτικό σφάλμα. Και το λέω αυτό για το επιχείρημα πίσω από την ιδέα αυτή. Ήταν ε, να γίνει καλύτερη η πολιτική μάχη για τη ΣΕΤΑ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι πολιτικό το σφάλμα, γιατί ήταν πολλές εθνικές κυβερνήσεις που δεν ήταν διατεθειμένες να ανοίξουν τη συζήτηση αυτή στο εσωτερικό τους για ένα πράγμα το οποίο ήταν σημαντικό, αλλά δεν ήταν έτοιμε να εκτεθούν σε δημόσιο διάλογο. Και έτσι δώσαν την πρωτοκαθεδρία στους λαϊκιστές. Και κάτι ακόμη που τροφοδοτεί του λαϊκιστές σε όλε τι χώρε αυτή τη στιγμή, είναι ότι λέμε πω πρέπει όλο και προς τώρα να ακούγεται τη φωνή των εθνικών κοινοβουλίων. Βεβαίω τα εθνικά κοινοβούλια εκπροσωπούν του πολίτε. αλλά και εμεί εκπροσωπούμε του πολίτε. Εγώ προσωπικώ εκπροσωπώ του πολίτε τη χώρα μου και υπάξια. εισάξια τουλάχιστον με οποιονδήποτε εθνικό βουλευτή της χώρας μου. Εάν λοιπόν μου λέτε ότι πρέπει για την εμπορική πολιτική, που είναι αρμοδιότητα αποκλειστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίε, πρέπει να ζητούμε τη γνώμη ενός Εθνικού Κοινοβουλίου, δεν δίνεται περισσότερη δύναμη σε αυτούς που προσπαθούν να αποδιαρθρώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο το σύστημα. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι έχω περάσει τον χρόνο. Αλλά είναι η ίδια κατάσταση, το ίδιο παιχνίδι και οι ίδιε κατευθύνσει. Εσεί βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φίγκλερ. Η κυρία Μόσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Υπογραμμίστηκε από πολλούς και συμμερίζομαι τις απόψεις τους ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνος λόγος των ανισοτήτων, έστω και αν αυτή την εικόνα δίνεται, δίνει γενικότερα. Ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ωφέλη της εμπορικής πολιτικής δεν έχουν διαμοιραστεί ισότιμα και υπάρχουν πολλοί που είναι χαμένοι από αυτή την υπόθεση. Όλο και περισσότερο προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε αυτές τις ανισότητες και λέγεται ότι πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανισότητες μέσω μέτρων που θα συνοδεύουν αυτές τις συμφωνίες προς όφελος των χαμένων για να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα της εμπορικής πολιτικής. Αλλά, και εδώ έχετε η ερώτησή μου, Πώς είναι δυνατόν σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα να μπορέσουμε εκ των προτέρων να ε, εντοπίσουμε τους τομείς, τους χώρους, τις γεωγραφικές ακόμη περιοχές που μπορεί να υποστούν κατά το μάλλον τις συνέπειε μια μιας εμπορικής συμφωνίας όταν βλέπουμε ότι οι μελέτε συνεπειών και πρέπει να γίνονται όλο και τώρα ε, δεν αρκούν τελικά για να καταγράψουν τις εξελίξεις για να προβλέψουν την πραγματικότητα και τα μέτρα που καλούμε να αναλάβουμε και επιπλέον πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα επιμέρους κράτη-μέλη στην υλοποίηση των μέτρων αυτών που θα επιτρέψουν την περιστολή των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη και για διαφοροποίηση. Αλλά και ανάγκη από πλευράς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν και να καθοδηγήσουν τις κυβερνήσεις για να υπάρξει από πλευράς των κρατών μελών άμεση και ενεργός παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν να στραφώ στους ε, διακεκριμένου μα ομιλητές, έχουμε λάβει και κάποιες ερωτήσεις από το Twitter και θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπέρτ Λάγκερ για να μας τι υποβάλει. Ναι, πολλές ερωτήσεις ε, τις έχω ομαδοποιήσει. Πρώτα προς τον κύριο Μπέρνερ. Οι μεγάλες διμερείς συμφωνίες θα υποβαθμίσουν ε, τις, τον, την, την ισχύ του ΠΟΕ Έπειτα, ποιε οι επιπτώσει των εμπορικών συμφωνιών είναι σχετικά περιορισμένε ο αντίκτυπο μάλλον. Μήπω θα ήταν ε, καλύτερο να εστιαστούμε σε πολυμερέ επίπεδο, ιδιαίτερα ε, σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στι διμερείς συμφωνίε γιατί μην παίρνουν τόσο χρόνο μέχρι να συναυθούν. Δεύτερον, είναι καλύτερο να μετακινούνται τα γεωργικά προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο αντί να ενισχύσουμε την περιφερειακή προστασία ή προστατευτισμό. Αυτό σε σχέση με την βιωσιμότητα και την οικονομική απόδοση. Και ε, Σεσίλια για σένα, για το εμπόριο που βασίζεται σε αξίες και για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιράν και ανθρώπινα δικαιώματα και διαπραγματεύσεις ΤΕΖΑ σε σχέση με την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης του Πακιστάν. So it is, uh, it is. Ο κύριος Βίνκλερ, δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν εγώ πρέπει να σας πω πως ίσως έχετε πέντε λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε. Πρώτα η Επίτροπος Αρμόδια για το Εμπορίο, η κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που νομίζω ότι απευθύνονται σε μένα. Αν δεν νομίζετε ότι απαντώ, να επανέλθετε, παρακαλώ έχει νόημα το να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά στις, στις συμφωνίες. Εμείς διαπραγματευόμαστε με την κυβέρνηση του ΙΟΝΙΠΑ για το τι μπορούμε να κάνουμε στο TTIP. Γι' αυτό το συμπεριλαμβάνουν στις διαπραγματεύσεις για το TPP. Έχει νόημα γιατί αν είναι σαφείς οι κανόνες και διαφανείς αυτό διευκολύνει το εμπόριο. Όμως η φοροδιαφυγή είναι πιο περίπλοκη για να μπει στις ε, εμπορικέ συμφωνίες. Υπάρχουν άλλα φόρα πιο κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν το θέμα, αν και αναγνωρίζω τον, την οργή των πολιτών για την φοροδιαφυγή, την ε, φοροαπάτη, Panama Papers και ούτω καθεξής. Για τις Φιλιππίνες, ναι, ανησυχούμε για πράγματα που γίνονται εκεί και θα, μάλιστα θα πάμε σε μερικές μέρες και ελπίζω πως οι αρχές των Φιλιππινών θα είναι συνεργάσιμες και θα σας πούμε τι έγινε. Για τους δασμούς, Στη ΣΥΠΑ είναι υποθετικό το ερώτημα. Ίσως ο φίλος μας από το ΠΟΕ έχει πιο συγκεκριμένες απόψεις. Είπατε κάτι τώρα για το εμπόριο. Το εμπόριο εδώ και δεκαετίες έχει αρμοδιότητα η Ένωση. Γι' αυτό έχει, έχουμε συνάψει 40 εμπορικές συμφωνίες σε διαφόρων επιπέδων και αυτό το έχουμε κάνει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαπραγματευτεί με την ισχύ ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια. Αν αυτή η αρμοδιότητα αφαιρεθεί, και καταλαβαίνω ότι κάποια κρατημέλη θέλουν να επανεθνικοποιήσουν κομμάτια ή ολόκληρη και την εμπορική πολιτική. Θα ήταν αυτό καταστροφικό για την Ένωση. Όχι γιατί εγώ θα μείνω χωρί δουλειά, γιατί εγώ μπορώ να βρω άλλη δουλειά, αλλά γιατί η ισχύ ολόκληρη εσωτερική αγορά είναι πολύ ελκυστική για του εταίρου μα και θα ήταν πολύ αρνητικό για τον πλούτο μα, για την ποιότητα των εμπορικών μα συμφωνιών και βεβαίω για ένα σωρό άλλους λόγους, εάν δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ως Ένωση. Είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Ε, τα κράτη-μέλη συμφωνούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει το θέμα τώρα το που ακριβώς είναι το όριο της εθνικής και της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και η Λισαβόνα δεν είναι σαφής γι' αυτό ακριβώς, αυτό πρέπει να το δεχτούμε και γι' αυτό και έχουμε στραφεί στο δικαστήριο με την υπόθεση της Σιγκαπούρης. Είναι ατυχές που η συμφωνία της Σιγκαπούρης είναι το σύμβολο αυτής της υπόθεσης, αλλά ελπίζουμε πως το δικαστήριο θα μας δώσει μια σαφήνεια και θα μπορέσουμε μετά να σχεδιάσουμε σχεδιάσουμε καταλήλως και την εμπορική συμφωνία. Αλλά και αυτό βέβαια εξαρτάται από την πολιτική στήριξη, γιατί κάποια κράτη-μέλη ισχυρίζονται ακόμα και πριν συμφωνήσουν με την εντολή ότι θα είναι μεικτή συμφωνία και τελικά εκείνοι αποφασίζουν. Αλλά ναι, πρέπει να το σκεφτούμε πραγματικά και θα γίνει η συζήτηση σχετικά ήδη την Παρασκευή όταν θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εμπορίου και θα αξιολογήσουν τα της ΣΕΤΑ και φυσικά κάποιοι εταίροι μας ρώτησαν μπορεί να συνάψει κανείς ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθείτε να είστε αξιόπιστος εταίρος μπορούμε να σας εμπιστευτούμε ότι θα, το, ότι θα την ε, υιοθετήσετε και εκεί αρχίζει, παίζει, αρχίζει ο ρόλος των κρατών μελών και των κοινοβουλίων. Γιατί τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν με την έννοια ότι να παρακολουθούν τη συζήτηση. Και αυτό το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι τα κράτη-μέλη μόλις εγκριθεί εντολή για διαπραγμάτευση με τη Διντάδη τη Δυναχώρα θα πρέπει να ανοίξουν το θέμα και στο κοινοβούλιο τους, να εξηγήσουν γιατί είναι καλό, γιατί είναι θετικό και να φέρουν και τις ερωτήσεις ε, εδώ ναι, ναι, να, υπάρχει λοιπόν συζήτηση μεταξύ όλων και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε ε, κάθε φορά να συμμετέχουν τόσο τα Εθνικά Κοινοβουλία όσο και η κοινωνία των πολιτών και οι διάφοροι φορείς ε, κρατικοί. Και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν εθνικές μήνυ ε, εκτιμήσεις αντικτύπου, μελέτες αντικτύπου, για να εντοπίσουν τις, τα ισχυρά σημεία αλλά και τις αδυναμίες, καθώς και τους τομείς κινδύνου σε κάθε χώρο σε κάθε χώρα, ώστε πριν να συναυθεί η συμφωνία να έχουν γίνει προσπάθειες άβληση των αρνητικών ίσως επιπτώσεων. Κάποιοι τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά, αλλά κάποιοι άλλοι καθόλου ώστε οι διάφορες πολιτικές για το πώ θα προστατευτούν οι δυνητικοί χαμένοι ε, να υπάρχουν ήδη. Το μέλλον του ΙΣΤΙΤΙΠ ήταν τελευταίο. Ποιος ξέρει συζητάμε τα τεχνικά ζητήματα με την σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε κάνει κάποιο πρόοδο. Θα πρέπει στο τέλος του έτους να αξιολογήσουμε την πρόοδο. Θα σας ενημερώσουμε και μετά βεβαίως θα υπάρξει μια, ένα διάλειμμα. Πόσο θα διαρκέσει εξαρτάται από την επόμενη κυβέρνηση να δούμε αν και κατά πόσο θα θελήσει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Ειλικρινά όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχει νόημα να υπάρχει συμφωνία εμπορική ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Πολλοί στην Ένωση αυτό το υποστηρίζουν και στη ΣΥΠΑ επίσης. Αλλά πότε θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει, δεν μπορώ να σας πω. Τέλος. Εσεί τώρα παριθμίσατε ένα σωρό ερωτήσεις οι εμπορικέ συμφωνίε δεν μπορούν από μόνο να λύσουν τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικά και όχι. Αλλά αν θα συνδυαστούν με πιο στρατηγική εξωτερική πολιτική όσον αφορά την ε, βοήθεια για το εμπόριο, την εξωτερική πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική και τα διάφορα εργαλεία συνεργασίας, Αναπτυξιακή συνεργασία. και έτσι προσπαθούμε να δουλεύουμε στην Κομισιόν, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και το εμπόριο θα παίξει το δικό του ρόλο. Θα, μπει και, θα μπουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα δίπλα με ε, ε ρήτρε για την βιώσιμη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Να δημιουργήσουμε πλατφόρμες για να μπορούμε να συζητήσουμε με τους εταίρους μας, να πιέσουμε ε, να υπάρχει και η δυνατότητα αναστολής αλλά σίγουρα να πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εντάσσονται στις αξίες. Δεν μπορούμε μόνοι μας να αλλάξουμε μια δικτατορία σε δημοκρατία μέσω μιας εμπορικής συμφωνίας, αλλά μπορούμε να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας. Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν σε μένα. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, πολλά διδάγματα μπορούμε να αποκαμίσουμε από τα τα πρόσφατα γεγονότα και θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Υπήρξατε η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Εμπορίου. Είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθετε εδώ στους κόλπους της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μπρούνερ. Ευχαριστώ. Μπράουνερ, συγγνώμη. Ο κύριος Φιέλνερ ρώτησε τι θα γίνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πιο σύγχρονη και πιο σε βάθος προσέγγισή της απομακρυνθεί από την υπόλοιπη κοινότητα του ΠΟΕ και παίξει ένα ρόλο πρωτοπόρου που ξεφεύγει. Τουλάχιστον έτσι κατανόησα την ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στον ΠΟΕ. Και επειδή εγώ είμαι Ευρωπαίος, είμαι, τόσο, είμαι ακόμα πιο ευχαριστημένος για τον ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου διότι βάζει και τις κατευθύνσεις σε πολλά θέματα και επιβάλλει τις τάσεις. Καμιά φορά με ιδέες που δεν ε, είναι ακόμα όριμες για τους καιρούς. Εμπόριο και επενδύσεις που χρειάστηκε, η πρόταση δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει το 2003, τώρα όμως επανέρχεται στην μέση έδραση. Κύριε Μάρτιν, ίσως να μην ήμουν απόλυτα σαφής. Μιλήσατε για ένα συμβιβασμό στον οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ήθελα να πω εγώ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμένει στις αρχές της και άρα κάνει μια θυσία με τις παρατεταμένης διαπραγματεύσει και όχι με ένα σύντομο αποτέλεσμα. Πέρασα πρόσφατα από το Χονγκ Κονγκ όπου μπόρεσα να ρωτήσω τον Μαλαισιανό Υπουργό Εμπορίου πώς και έχει συμφωνία Free Trade Agreement με την Ιαπωνία και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεξέφυγε στην απάντησή του, ωστόσο εγώ θεωρώ ότι η Ιαπωνία δεν φάνηκε να βασίζει τη στάση της τόσο πολύ σε αξίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό που λέω είναι ότι δεν συμβιβάζεται. δεν συγχωρείτε λέει ο κύριος Μάρτιν. Το κατάλαβα πολύ καλά αυτό που, εξή, εξηγήσατε. Η ερώτησή μου ήταν πέραν αυτού. Δεν λέω ότι ε, πρέπει οι διαπραγματεύσεις να είναι παρατεταμένες λόγω διαδικασιών. Α, μάλιστα. Από αυτού δεν έχω σχόλιο, λέει ο κ. Τώρα θα ήθελα να σας πω ε, μια ιστορία ε, εκτός αρμοδιοτήτων μου, αλλά υποκύπτω στον πειρασμό. Στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα, ελπίζω να μην προσβάλλω κανένα, ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου συναντάται με τον Πρωθυπουργό της Κίνας και συζητούν. Και στο τέλος της συζητήσεως ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου λέει «Καλά κάναμε και συνομιλήσαμε διότι μαζί εκπροσωπούμε 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και το απαντά ο Κινέζος Πρωθυπουργός και να φύγετε εσεί, εγώ εξακολουθώ να εκπροσωπώ 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Οποιοδήποτε και αν ήρθε από την Ευρώπη να συνομιλήσει με τον Κινέζο Πρωθυπουργό και να φύγει, <laughs> εξακολουθεί ο Κινέζο Πρωθυπουργό να εκπροσωπεί 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Το μήνυμά μου είναι ότι σοβαρά θα μας πάρουν μονάχα ως Ευρωπαίους, ως ενωμένους Ευρωπαίους. Με συγχωρείτε, είπα εγώ, μίλησα στο πρώτο πληθυντικό, ε, αλλά εγώ είμαι του ΠΟΕ βεβαίω, έτσι. Άρα, με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο μόνο ενωμένη, όχι ποτέ μια χώρα μόνη της. Και αυτό είναι ιδιαίτερα καθαρό στον ΠΟΕ, όπου όταν κάποιος θέλει να επιτύχει κάτι, πρέπει να διαμορφώσει συμμαχίες, να βρει ομάδες που θα τον στηρίξουν. Άκουσα και την ερώτηση εάν οι περιφερειακές ε, εμπορικές συμφωνίες θα υπονομεύσουν το έργο του ΠΟΕ. Όχι. Όταν μπαίνετε σε περιφερειακές εμπορικές προσυμφωνίες, επιλέγετε έναν εταίρο και όταν είστε επιτυχημένος για να επιτύχετε δηλαδή πρέπει να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις αντιστάσεις και στις δύο χώρες που συμμετέχουν στην ε, συμφωνία. Και υπάρχουν πολλές συμφωνίες ελευθέρου εμπόριου, free trade agreements, διαφόρων εταίρων, όπου ε, από τη μια μεριά ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εταίρος Χ από την άλλη και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλος εταίρος ε, Ψ από την άλλη μεριά και αυτό που κάνετε είναι σε ένα διμερές επίπεδο απαλύνετε τις αντιστάσεις. Αυτό σας επιτρέπει να έλθετε στο πολυμερές επίπεδο και να καταλήξετε πολυμερός πλέον σε μια επιτυχή λύση. Κάτι που είναι σημαντικό και πως τόσο αποτελεί ένα φραγμό για την ώρα είναι αυτοί οι κανόνες προέλευσης. Μιλήσαμε για παγκόσμιες ε, ε, αλυσίδες αξιών. Όταν η αλυσίδα είναι πολύ μακρά και κάθε φορά πρέπει να σέβεστε τους κανόνες ε, της προέλευσης για να εποφελείστε από τις προτιμήσεις, καθίσατε τελικώς αδύνατον να ισχύσουν αυτές οι εμπορικές συμφωνίες. Αυτές ήταν οι απαντήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, λέει ο κύριος Βίνκλερ που διευθύνει τη συζήτηση και θα δώσω το λόγο τώρα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, τον κύριο Φρανκς. Θα είμαι σύντομο. Εάν παραλείψω να απαντήσω σε κάποια ερώτησή σας, πιάστε με μετά και πέστε τα μου διμερός. Πολύ ευχαρίστω. Σχολιάζω πρώτα κάποιες παρατηρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφενός να φορτώνουμε όλα τα κακά στις εμπορικές συμφωνίες. Καμιά φορά οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να είναι υπεύθυνε για κάποια κακά πράγματα, αλλά μην τις φορτώνετε όλα. Και από την άλλη μεριά, μην αναμένετε οι εμπορικές συμφωνίες να λύσουν όλα τα προβλήματα. Πρέπει να τις δούμε από τη σωστή προοπτική. Εάν υπάρχει πρόβλημα, για παράδειγμα, στις συνθήκες εργασίας και στους μισθούς, πρέπει να επιληθούν αυτά τα προβλήματα πρώτα. Μη προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο εργαλείο παίρνοντα από την πίσω πόρτα. Σωστό είναι να ληφθούν υπόψη βεβαίω πράγματα όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκε εργασία, περιβαλλοντικά και ούτω καθεξή. αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ασφαλώ και πρέπει να σα απασχολήσουν. Όμω να χρησιμοποιείτε το όχημα των εμπορικών συμφωνιών για να αντιμετωπίσετε όλε αυτέ τι ανησυχίε, στην πραγματικότητα φορτώνεται το εργαλείο αυτό πάρα, πάρα πολύ. Είναι σωστό να χρησιμοποιηθούν τα σωστά εργαλεία για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά το όφελος και το κόστος του εμπορίου. Μια διευκρίνηση μετά από τα σχόλια που έγιναν εδώ για κερδισμένους και χαμένους. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό ότι υπάρχουν πιο πολλοί χαμένοι από κερδισμένους από τις εμπορικές συμφωνίες. Κάθε ένας που αγοράζει ένα τηλέφωνο, ένα ρολόι, ε, ένα ρούχο, εποφελείται από το εμπορίο. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τούτο εδώ το τηλέφωνο θα μπορούσε να κοστίζει εκατοντάδε ευρώ περισσότερα εάν δεν υπήρχε το παγκόσμιο εμπόριο. Οι άνθρωποι όμω που χάνουν τι δουλειέ του λόγω των εμπορικών συμφωνιών γνωρίζουν συχνά για ποιο λόγο έχασαν τι δουλειέ του. Και όπω είπαν και κάποια άλλα σχόλια, συχνά φορτώνουμε στο εμπόριο την απώλεια θέσεων απασχολήσεως. Όχι, δεν είναι το εμπόριο ο φταίχτης. Είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι η αλλαγή της τεχνολογίας. Συχνά, ωστόσο, είναι η εικόνα πιο συγκεκριμένη. Εάν, ωστόσο, εγκαταλείψουμε το διεθνές εμπόριο, τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει. Αν μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα σκεφτείτε χώρες οι οποίες το 1950, 60, 70 έβαλαν προστατευτικούς φραγμούς. Τελικώς αυτές οι χώρες υπέστησαν σημαντικές ζημίες. Αν δείτε τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοιχτές χώρες με πολλές εξαγωγές, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, φαίνεται καθαρά ότι αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα από αυτές οι οποίες ασκούν ένα προστατευτισμό. Μπορούμε να φανταστούμε την Κίνα να ε, μπορεί να άρει ένα δισεκατο... να σηκώσει ένα δισεκατομμύριο κατοίκους πάνω από το επίπεδο της φτώχειας χωρίς ε, τις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και να έρθω και σε ορισμένα άλλα πολυμερής έναντι περιφερειακών ε, εμπορικών συμφωνιών. Βέβαια, αυτά είναι, οι συμφωνίες αυτές είναι καλές, δεν παρεμβαίνουν στον γύρο της Ντόχα, όμως εξακολουθούν να είναι σημαντικές να προωθηθούν στο παγκόσμιο επίπεδο οι πολυμερείς συμφωνίες. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα στη σύγκριση τοπικής απέναντι στην περιφερειακή παραγωγή. Εφόσον θέλετε αγοράζετε τοπικά. Κάντε το. Ενισχύστε τις τοπικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τις τοπικές βιομηχανίες και το καθεξής. Δεύτερο, πρέπει να φροντίσουμε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και η τοπική και η διεθνής παραγωγή πρέπει να περιλάβει στην, στις τιμές και τα εξωτερικά στοιχεία όπως προστασία περιβάλλοντος και το καθεξής. Και εφόσον το κάνουν αυτό τότε θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ε, ποιο είναι το πραγματικό κόστο. Για παράδειγμα, το να πάτε με το αυτοκίνητο κάποια χιλιόμετρα για να αγοράσετε από μια κοντινή αγροτική εκμετάλλευση μπορεί περιβαλλοντικά να έχει μεγαλύτερο κόστο από το να έρθει ένα τεράστιο πλοίο φορτωμένο μαζικά εμπορεύματα και να τα βιάσει το λιμάνι. Α, κάνω και κάποια τελευταία σχόλια τα προβλήματα τα, του είδους που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο διαβαίνουν τα εθνικά σύνορα όλο και περισσότερο και ως αποτέλεσμα και οι απαντήσεις στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να διαβαίνουν τα εθνικά σύνορα είτε πρόκειται για εμπόριο, είτε πρόκειται για περιβάλλον, είτε πρόκειται για άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε από τον παρακαλώ, είναι ο τελευταίος. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα το σχετικό με τη διαφάνεια εξορισμού. Όταν έχουμε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη προβλεψιμότητα, βεβαιότητα, προφανώς υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για περιορισμό των ε, κινδύνων, ή πιθανότητων, διαφθοράς, αντίξεων, συνεπειών κτλ. Ενώ όταν είναι... Και έτσι όταν είναι διαφανής η κατάσταση, είναι γνωστή δηλαδή οι κανόνες του παιχνιδιού, είναι πιο δύσκολο και κάποια στελέχη να δωροδοκηθούν. Θα έλεγα επίσης ότι αν δεν υπάρχουν δυνατότητες ε, άλλες, ε, όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε την παγκοσμιοποίηση, η λύση είναι να κάνει καλύτερες, ε, καλύτερη νομοθεσία στο εσωτερικό της χώρας του για τη γεωργία και όλα αυτά. Το να έχει την επιλογή ο καταναλωτής να αποφασίζει τι θα αγοράσει, να αγοράζει με τα τοπικά προϊόντα χωρίς να είναι υποχρεωμένος, επειδή θα είναι κλειστές οι αγορές, είναι βέβαια λογικό. Αλλά εάν ε, ε, επιβληθεί περισσότερο προστατευτισμό στην γεωργία Φερρυπίν, θα γίνουν πιο πτυτικέ οι τιμές, πιο ασταθείς, θα αυξηθούν εν τέλει και άρα πιο πολλοί θα είναι αυτοί που θα μένουν ιστικοί στον κόσμο. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Το ίδιο ισχύει και για το περιβάλλον και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας απασχολεί κοινωνικέ κοινωνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Και κάτι ακόμη που επισημάνθηκε, ότι η πρόσθετη δυνατότητα επιλογής ή οι τιμές, οι πιο χαμηλές τιμές που προκύπτουν επειδή είναι καλύτερος ο ανταγωνισμός ή γιατί τα ιδεώδη, τα αγαθά, οι υπηρεσίες ε, ε διασχίζουν σύνορα. Αν δεν το θέλει κανείς αυτό, ε, πρέπει να κλείσει αγορές. Αν θέλει όμως ανάπτυξη, καλύτερες θέσεις εργασίας, πρέπει να ανοίξει τις αγορές του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμέσως θα φέρουν τα ωφέλη τους οι ανοιχτές αγορές. Αυτό προσπαθούσα να πω και στην αρχή της ομιλίας μου ότι είναι αναμφισβήτητα τα ωφέλη από το ρεύμα των αγορών, αλλά το ότι θα είναι τα ωφέλη αυτά ε, ε, στη διάθεση των πάντων δεν είναι δεδομένο εξ αρχής. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν να συμβαίνει τώρα δεν είναι η αποτυχία της παγκοσμιοποίησης, αλλά η αποτυχία των εσωτερικών πολιτικών που δεν ε, δίνουν λύσεις σε θέματα αναδιαμονωμής αυτού του πλούτου. Ίσως ε, δεν κάνουμε αρκετά καλή πολιτική ε, δημοσιονομική, διαρθρωτική. Σας ευχαριστώ πολύ, Ίσως. λέει ο Πρόεδρος. Δυστυχώ έχουμε εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο αυτό το κομμάτι τη συζήτηση. Δεν μπορώ να δώσω, λοιπόν, να δώσω το λόγο σε άλλου ε, συναδέλφου, αλλά αν μου επιτρέψετε θα πω μόνο δύο λέξεις, κυριολεκτικά δύο λέξει. Better together, καλύτερα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εσύ Πρόεδρε σας ε, παραδίδω το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ, εξαιρετική δουλειά κύριε Βίνκλερ, ευχαριστώ τους ομιλητές και καλό τους ομιλητές για το δεύτερο γύρο να έρθουν ε, στο Προεδρείο για να συνεχίσουμε την επικοδομητική πιστεύω αυτή συζήτηση. Thank you. Thank you very I Hello. No, So we had, she's here. Tiziana is coming? No. So, ladies and gentlemen, now we are coming to our second... Αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνουμε στο δεύτερο γύρο των συζητήσεων ιδιαίτερα στη συζήτηση που αφορά εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο και τη ΣΕΤΑ, που απασχόλησε και κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης συγκεκριμένα, έγιναν διαδηλώσεις, έγινε δημοψήφισμα στις κάτω χώρες, κατά της συμφωνίας ε, ελεύθερο μπορεί με την Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες είχαμε ζητήματα και σε σχέση με το, οι εμπορικές αλλαγέ με τι ΗΠΑ και την νομιμότητα αυτών των συμφωνιών. Αναζήτηση της εμπιστοσύνης, νομιμοποίησης ε, αναζήτηση μια νομιμοποίηση για το διεθνέ εμπόριο και νομίζω ότι έρχεται την καταλληλότερη δυνατή στιγμή. Οι ομιλητέ μας είναι εδώ νομίζω. Ε, more, more than the first one. So, um, the experts we have here... Έχουμε λοιπόν, λοιπόν εδώ τον κύριο Ιωάκιμ Χάιτα, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της UNCTAD, του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Εθνών. Έχουμε τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου, τον κύριο Σαντα Καταρίνα της Oxfam Magazine du Monde και τον κύριο Πολ Τουέντιν, επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Με τη σειρά που ακούσετε τα ονόματα θα γίνουν και οι παρεμβάσει. Και έτσι παρακαλώ τον κύριο Ιωάχιμ Ράιτερ να κάνει τις τοποθετήσεις του στο θέμα Quest Forest. Περισσότερη εμπιστοσύνη λοιπόν και νομοποίηση για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κύριο Ράιτερ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ. Ε, είναι άμεσος, άμεση συνάφεια της θεματολογίας των δύο ομάδων ομιλητών, των δύο πάνελ και άλλωστε έθιξαν το ζήτημα της νομιμοποίησης οι προηγούμενοι ομιλητές σε πολλές περιστάσεις. Εγώ θα ήθελα να πείσω το θέμα αυτό σε τρεις παραμέτρους. Καταρχάς υπάρχει νομοποίηση αυτή καθεαυτή για το διεθνές εμπόριο, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε νομοποίηση ως προς την εμπορική πολιτική και τι νομοποίηση έχουμε σε σχέση με την χάραξη πολιτικής για το εμπόριο. Τρία θέματα, αλλά δεν χρειάζεται να τα πραγματευτούμε χωριστά. Ακούστηκε λοιπόν νωρίτερα ότι αναπτύσσεται με πολύ βραδείς ρυθμούς ε, το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών. Αυτό ισχύει για όλους, αλλά ίσως να είδατε και το ανακοινώθεν της UBS ε, ότι οι υπηρεσίες, ε, οι συναλλαγές σε υπηρεσίες έχουν εξαπλάσια ανάπτυξη από αυτές των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών σε προϊόντα και αυτό σημαίνει ότι περνούμε σε μια κοινωνία με ιδιαίτερη έφαση στις υπηρεσίες, στην ε, μίσθωση προϊόντων βιομηχανικών και, στις χρηματοπιστωτικές, και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε εάν αυτές οι εξελίξεις μπορούν να ε, στηρίξουν τις αυξήσεις ε, τις μισθολογικές που είδαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Υπάρχουν σημαντικές πιέσεις αυτή τη στιγμή και άρα όχι μόνο στους μισθούς αλλά και στην ανάπτυξη ως εκ τούτου. Προκλήσεις λοιπόν, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Η εμπορική πολιτική. Η εμπορική πολιτική πολλών κρατών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι εν γέννη η εμπορική πολιτική ήταν πολιτική ανέκαθεν που αντιμετώπιζε σημαντικές προκλήσεις τώρα που είναι όλο και πιο ενωμένε μεταξύ τους και αλληλένδετε οι οικονομίες μας. βεβαίω είναι και μεγαλύτερες οι προκλήσεις και τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα θυμάστε ίσως ε, τις ε, τεράστιες διαδηλώσεις κατά του ΠΟΕ πριν από 15-20 χρόνια στο Σιάτλ παραδείγματι. Εγώ χρειάστηκε να εμφανιστώ ενώπιον του Σουηδικού Κοινοβουλίου την εποχή εκείνη με τα τότε καθήκοντά μου να υπερασπιστώ τη Σουηδική πολιτική για το εμπόριο. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το εμπόριο αλλά και με άλλα ζητήματα. Έχουμε όλο και περισσότερο όγκο προβλημάτων ε, σε σχέση και με τα εσωτερικά μέτρα και τα διασυνοριακά δεδομένα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση ε, ηλεκτρονικών δεδομένων. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν που μπαίνουν μέσα στην εμπορική πολιτική δίνουν και, δεύτερους, και νέους διαφορετικούς στόχους και πεδία δράσεως για την εμπορική πολιτική που δεν είναι απαραίτητα πεδία δράσεως ευχερούς για την πολιτική του εμπορίου. Δεν είναι κάτι δηλαδή, στο οποίο έχουμε συνηθίσει να δρούμε όταν κάνουμε μια συμφωνία εμπορικών συναλλαγών, ε, ε, αγοραπολισίες προϊόντων κτλ. Και πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα του infinite governance, της απεριόριστης ή απέραντης διακυβέρνησης. Το διαδίκτυο λοιπόν έχει τελείως διαφορετικές και τεράστιες θα έλεγα δυνατότητες από αυτές του ε, εμπορίου πρέπει να μπορέσουν να συνενωθούν και να συνδυαστούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πάνω από όλα ότι έχουμε ε, ένα τεράστιο όγκο προκλήσεων μπροστά μα, αλλά ταυτόχρονα το έχουμε και την ε, αποδεδειγμένη δυνατότητα από το παρελθόν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι δυνατότητε. Όπω όταν είχαμε τι συναλλαγέ σε προϊόντα, σε υπηρεσίε μέσα από τον ΠΟΕ, είχαμε μπορέσει να δώσουμε απαντήσει στα προβλήματα στη δεκαετία του 90. Η εμπορική πολιτική λοιπόν να μην καν, μπορεί να μην είναι καν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, μεγάλο πρόβλημα, ναι, μεγάλε προκλήσει. Πρέπει με ταπεινότητα να στραφούμε και να πούμε στη εθνική κοινότητα ότι δεν έχουμε όλε τι απαντήσει έτοιμε. Και τώρα έχουμε την γενική χάραξη πολιτική για το εμπόριο και ζητώ συγγνώμη που θα είμαι ομός. Οι γενικότερες πολιτικές του εμπόριου είναι αχταρμάς. Και για διάφορους λόγους. Δεν μιλούμε για πυρηνική φυσική εδώ. Τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι με την εμπορική πολιτική βλέπουμε να γίνεται να μετατρέπεται σε ένα θέμα το οποίο ε, εξειδικεύεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή κάποιος ασχολείται μόνο με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του anti-dumping, μόνο με ένα συγκεκριμένο κομμάτι των εμπορικών φραγμών. Και όμως αντίστροφα ε, αντίθετα το εμπόριο είναι διανεμητικό εκ της φύσεώς του. Αυτή είναι η φύση του και ως εκ τούτου δεν αρκεί να προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέλημα το οποίο μπορεί να αισθάνεται η κοινωνία ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με την ανάπτυξη ενός τομέα του εμπορίου. Άρα γύρεται το ζήτημα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε συνένεση εθνικό επίπεδο για το εμπόριο, αλλά και πώς να ε, προχωρήσουμε μέσα σε μια ασφαλή ζώνη, μέσα και έξω από την εμπορική πολιτική που να επιτρέπει την διανεμητική λειτουργία του εμπορίου. Και ξέρω ότι δεν ε, έχω περιθώριο να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να είμαι πολύ τόσο ξεκάθαρος πως δεν πιστεύω ότι οι λύσεις που μπορούν να συνδυάζονται με πολιτική για το εμπόριο είναι αυτές οι οποίες μπορούν να λύσουν τα πολιτικά προβλήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή χάρη στο εμπόριο να δώσουμε απαντήσεις σε ανησυχίες πολιτικής φύσεως και μελήματα ή αγωνίες που επικρατούν και που μάλιστα πρέπει να σας πω επικρατούν στον πλούσιο κόσμο. Επίσης δεν νομίζω ότι αποτελεί λύση να δώσουμε ε, να, δώσουμε λύσεις σε διαδικασίες με διαδικοστικά βήματα. Δεν θέλει κανείς να ακούσει δηλαδή ότι θα γίνει άλλο ένας γύρος ε, διαλόγου. Θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις για την θέση εργασίας που αναζητά. Και γενικά ακούμε ότι οι αρμοδιότητες για την, ευρωπαϊκή, για την εμπορική πολιτική είναι ομοσπονδιακή, ενώ η πραγματική απάντηση για τα μελήματα των πολιτών θα δοθεί από εθνικά, εσωτερικά μέσα. Άρα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί κάπου για να πει τι είδους κοινέ απαντήσεις μπορούν να χορηγηθούν, μπορούν να δοθούν στον πολίτη με την εφαρμογή αυτού του ομοσπονδιακού μέσου που είναι το εμπόριο μέσα από την εθνική πολιτική. Όπως είπε ο κύριος Σάσο από τον ΩΣΑ, κοινωνική προστασία, αναδιανομή. Συγκεκριμένο παράδειγμα, το σύστημα προσαρμογής, η υποστήριξη στην προσαρμογή στο εμπόριο, ε, είναι ένα δολάριο στα 250 στα 2.500 δολάρια ε, μισθό. Δηλαδή είναι 0,004% επί του εισοδήματο του καθενός. Είναι ένα πυροελάχιστο κομμάτι σε μια οικονομία των 13 εκατομμυρίων σε ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσοστό μη βιώσιμο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Επομένω πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Και άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μια μέθοδο να δώσουμε απαντήσεις ε, πολιτικής σχετικής με το εμπόριο, που θα δίνει απαντήσεις στα προβλήματα, αλλά και θα μεγιστοποιεί τα ωφέλη. Πραγματική εμπορική πολιτική δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη σοβαρά το ζήτημα και του ανταγωνισμού, αλλά και της προστασίας του καταναλωτή. Ιδάλλως, τα ωφέλη του εμπορίου, πολλά, ανεγνωρισμένα, και τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, θα περιοριστούν μόνο σε πολύ ε, ολίγους. Άρα πρέπει να ενισχυθούν και οι κανόνες για την προσοχή του καταναλωτή και οι κανόνες για τον ανταγωνισμό και ήδη πολλέ χώρε το πράττουν αυτό. Και, άλλα, και άλλοι τομεί όμως πολιτικής. Πολιτική για την εκπαίδευση παραδείγματι που έχει τεράστια σημασία. Καταλήγω στο ότι δεν υπάρχει επιλογή άλλη από την κανονιστική ρυθμιστική συνεργασία. Το είπε κάποιο νωρίτερα ότι έχουμε ζητήματα διασυνοριακά, υπερσυνοριακά, τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ο καθένα χωριστά στα ιστορικά του σύνορα. Επίση, έχουμε όλο και μεγαλύτερη ζήτηση από τι διάφορε χώρε, ρυθμιστική προσέγγιση, παραδείγματι, που ε, ζητούν και οι χώρε Αφρική για να αντιμετωπίσουν τι δυσμενεί συνέπειε του εμπορίου. Ναι, βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική εμπορίου με βάση την αξία, αλλά μην προσπαθήσει να επιβάλλει τους κανόνες της σαν να ήταν ιεροκήρυκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα αυτό όταν προβαίνει κανείς σε συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με, με έναν εταίρο. Και αυτός περιμένει ότι θα τον ακούσει, ότι θα ακουστεί η φωνή του, ότι θα εκφράσει τις δικές του ανησυχίες και επιθυμίες. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Η ανάπτυξη της ζήτησης για βιώσιμα προϊόντα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή από ό,τι εκδηλώνεται στις πλούσιες χώρες. Γι' αυτό βλέπετε όλο και περισσότερο να αναπτύσσονται πρότυπα και προδιαγραφές για τέτοιου είδους προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχει πεδίο ως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνεργασία έχετε δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή τους με κηρύγματα. Πρέπει να συνεργαστεί. Δύο λόγια ακόμα για να κλείσω. Η διατήρηση του status quo δεν αποτελεί τίποτα άλλο από οπισθοδρόμηση, γιατί οι υπόλοιπε περιοχές του κόσμου προχωρούν. Δεν θα κάτσει κανείς να περιμένει να δει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ. Όλο και λιγότερα είναι τα ερωτηματικά ε, σε σχέση με την πολιτική για το εμπόριο που αναπτύσσουν οι υπόλοιπε ζώνες του κόσμου. Θα συνεχίσουν, θα έχουν μεγάλα δίκτυα των μεταφορών, όπως ε, έχει προχωρήσει η Κίνα σε τεράστιες ε, λωρίδες μεταφοράς ε, ε, προϊόντων, ανάπτυξη του ΑΕΠ και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αφήσει η Ευρώπη να περάσουν δίπλα της. Η μόνη λύση λοιπόν είναι η συνεργασία. Πρόεδρος Λάγκε, ευχαριστώ πολύ για τον ανοιχτό τρόπο που μιλήσατε. Γκονζάλες τώρα, γνωστός εδώ στις Βρυξέλλες, του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στις δημοκρατικές κοινωνίες οι ανοιχτές αγορές βασίζονται στην συνένεση της κοινωνίας. Αυτή η συνένεση της κοινωνίας σε πολλές ε, σημερινές κοινωνίες έχει γίνει πολύ εύθραυστη. Πρόκειται για κρίση νομιμοποίησης και είναι και ατυχής αλλά και κατανοητή. Και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και δύο πλευρές του προβλήματος. Γιατί είναι ατυχής διότι πρόκειται για ανοιχτές αγορές που μας, αυτές μας βοήθησαν να βγάλουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους από την φτώχεια, από την ακρότατη φτώχεια. Ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, ξαναλέω. Δεν είναι και κανένα μικρό κατόρθωμα. Η εξωτερική ζήτηση είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για να μεταμορφωθούν οικονομίες που στο παρελθόν βασίζονταν σε χαμηλές παραγωγικότητες. Αυτή η μεταμόρφωση, αυτός ο μετασχηματισμός είναι που βλέπουμε σήμερα στην Κένια, στο Βιετνάμ, στον Ισημερινό του Εκουαδόρ δηλαδή, λίγες χώρες αναφέρω, αλλά παίρνω από διαφορετικές υπήρους για να σας δώσω μια γεύση, και το τι γίνεται και στην Ευρώπη. Αν θυμηθώ το γερμανικό οικονομικό θαύμα που δεν θα είχε γίνει δυνατό εάν δεν ε, είχε βασιστεί αυτή η, αυτός ο μετασχηματισμός στην εξωτερική διάσταση, εξωτερική ζήτηση. Είναι ατυχές επίσης διότι αυτές οι οικονομίες που μας έδωσαν μεγάλη δυνατότητα συμμετοχής, άνοιγμα των επιλογών των καταναλωτών, κέρδη στην παραγωγικότητα, όμως ταυτόχρονα είναι και κατανοητή αυτή η έλλειψη συνένεσης, διότι οι επιχειρηματικές ελίτ και οι πολιτικοί δεν πρόσεξαν, πάντως το πρόσεξαν επαρκώς, το γεγονός ότι το άνοιγμα των αγορών θα έβλαπτε κιόλας μέρη του οικονομικού μας ιστού και περί αυτό πρόκειται. Έστω και αν συνολικά ε, είμαστε σε καλύτερη θέση, πάντως αυτό είναι που έρχεται τώρα και μας στοιχιώνει. Όταν δηλαδή το μικρό τράκαρε πάνω στο μάκρο. Δηλαδή στο μακροοικονομικό επίπεδο είμαστε καλύτερα, όμως η πραγματικότητα είναι ότι στο μικροοικονομικό επίπεδο υπάρχει πολύ μεγάλη δυστυχία. Είναι κατανοητό επίσης, διότι το εμπόριο έγινε το απτό σύμβολο των οικονομικών αλλαγών που διερχόμεθα, ακόμη και αν, αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, δεν είναι το εμπόριο εκείνο που θα πρέπει να μας ανησυχεί, Πάντως ε, δεν είναι εκείνο που θα πρέπει να μας ανισχύει τόσο πολύ. Ε, είναι το φάσμα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία που δυστυχώς δεν υπακούει σε δημοψηφίσματα, ούτε σε διαδηλώσεις, ούτε σε κοινοβουλευτικές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, που ωστόσο από την άλλη μεριά η τεχνολογία δίνει τεράστια δύναμη στο, στη βάση της πυραμίδας οδηγεί όμως και σε μεγάλες ταχύτατες ανατροπές στον οικονομικό ιστό. Άρα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στο πόσα φορτώνουμε στην πλάτη του εμπορίου και να ψάξουμε να βρούμε που πραγματικά βρίσκεται το πρόβλημα, να μην πυροβολούμε και τους αθώους. Άρα τα προβλήματα δεν λύνονται με εμπορική διπλωματία περισσότερο με εγχώριες οικονομικές και εμπορικές πολιτικές και βεβαίως οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κοινωνικές πολιτικές τους τα κατάφεραν καλά μέχρι τώρα να απαλύνουν την φτώχεια των ανθρώπων που σήμερα όμως οι προσπάθειες αυτές δεν επαρκούν πλέον. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό ε, συμβόλαιο και εδώ στην Ευρώπη. Εδώ όμως η διάκριση δεν είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, είναι ανάμεσα στις ανοιχτές και στις κλειστές κοινωνίες. Κοινωνίες οι οποίες δίνουν δύναμη στον άνθρωπο, στο άτομο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, αυτές δηλαδή τις οποίες προωθεί με μεγάλη ταχύτητα η τεχνολογία, αυτή η προετοιμασία στην προσαρμογή στις νέες ευκαιρίες επίσης που δημιουργούνται από την τεχνολογία στις πτυχέ εκείνες που δεν βοηθούν αυτή την προσαρμογή. Δεν θα μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το εμπόριο, έτσι. Ε, σας καθησυχάζω. Όλα αυτά έχουν σχέση και με το εμπόριο. Στο κάτω-κάτω εδώ Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου είσαστε. Πρώτον, λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι η φραγμή στο εμπόριο στον 21ο αιώνα είναι ρυθμιστικού χαρακτήρα. Ρυθμιστικός χαρακτήρας σημαίνει προκειμένου ποιότητα του εμπορίου και όχι ποσότητα. Η ποιότητα του εμπορίου έχει επίσης σχέση, όπως ακούσαμε και από τον Ιωακίμ Ράιτερ προηγουμένως, από την ασφάλεια μέχρι την προφύλαξη, μέχρι την ιδιωτική σφαίρα και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό χρειάζεται να διαφυλαχθεί το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν νομοθετικά. Δεύτερο, για να μπορέσει να αποδώσει το εμπόριο στον 21ο αιώνα πρέπει να είναι ανοιχτό, inclusive. Με έχετε ακούσει επαρκώ μέχρι ναυτίας λαμπίν το ξαναπώ λοιπόν, αρκεί να πω ότι 95% του οικονομικού ιστού κάθε μια από τι χώρε σα είναι οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Φροντίδα λοιπόν να φέρουμε τι νομοθετικέ ρυθμίσει κοντύτερα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει κοντύτερα στι ευκαιρίε που ανοίγει το εμπόριο. Αυτά είναι ουσιώδη πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμπόριο. Είμαστε, είσαστε εδώ, Επιτροπή Ίντα. Ανοιχτό εμπόριο σημαίνει ότι εν τέλει και οι γυναίκες θα μπουν στο διεθνές εμπόριο που τώρα ο ρόλος τους είναι πολύ μικρότερος από ό,τι των ανδρών. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πολιτικές. Αυτά δεν ισχύουν μοναχά για τις προηγουμένες οικονομίες, ισχύουν και για κάτι που θα πρέπει να σκέπτεστε εσείς για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου εξακολουθούμε να έχουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Τέλος, το εμπόριο πρέπει να μπει πιο ορατά στην υπηρεσία της αηφορίας, της βιωσιμότητας στο κάτω της γραφής Ευρωπαϊκή Ένωση. Είσαστε πρωταθλητές δηλαδή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του περιβάλλοντος, ωστόσο μην τα λησμονείτε. Ένα μέγα μέρος για να γίνει πιο ανοιχτή και πιο βιώσιμη η εμπορική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, όλες αυτές οι προσπάθειες δεν αρκούν. Οι εμπορικές πολιτικές πρέπει να συγχρονιστούν καλύτερα με τις ε, ε, εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το αποτέλεσμα στην διανομή του εμπορίου. Κάτι που δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Έχει σχέση με την εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την απόκτηση δεξιοτήτων, μια ενεργό πολιτική της αγοράς εργασίας και εν τέλει, γιατί όχι, και με ένα παγκόσμιο βασικό εισόδημα με πολιτικές καινοτομίας, με φορολόγηση. Και μιας και μιλούμε για φορολόγηση, έχει σχέση και με τη διεθνή συνεργασία για την μείωση της εταιρική φοροαποφυγής, που επίσης υπονομεύει τις δυνατότητές μας να ασκήσουμε ορθές εμπορικές πολιτικές. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε παραδείγματα χωρών που διατήρησαν ανοιχτές τις αγορές τους, που εφήρμοσαν πολιτικές και έχετε επίσης και χώρες με ανοιχτές αγορές και με λιγότερο λεπτομερείς και προηγμένες κοινωνικές πολιτικές. Εσείς θα διαλέξετε ποια παραδείγματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Δεν είναι δικός μου ρόλος να σας τα υποδείξω. Κατά τη γνώμη μου, η προκλήση που αντιμετωπίζετε σήμερα δεν είναι να διαλέξετε ανάμεσα σε ανοιχτές ή σε κλειστές αγορές. Δεν έχετε καν αυτή την επιλογή λόγω του φάσματος της τεχνολογίας. Όποιος από εσά θεωρεί ότι μπορεί να κλείσει την αγορά του και να προστατεύσει τους πολίτες του, sorry, δεν είναι δυνατόν. Η τεχνολογία δεν σας το επιτρέψει. Η επιλογή σας λοιπόν είναι ανάμεσα σε ανοιχτές αγορές και ενεργές πολιτικές που θα δώσουν τη δύναμη στο άτομο να προσαρμοστεί, είτε σε ανοιχτές αγορές χωρίς δίκαιη κατανομή αναμένω να δω τι θα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τι επόμενε εβδομάδε, διότι αυτό για μένα θα είναι το απότατο τεστ, η απότατη δοκιμασία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μπλάγκε. Κάποιε φορέ. ε, δεν ε, θέλω και πολύ να δω τέτοιες, ε, τέτοιες ε, δοκιμές, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εμείς συμμετείχαμε και ε, στον καθορισμό της εμπορικής εντολής. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για την εμπορική πολιτική. Έχει βελτιωθεί. Κοιτάξτε, έχω μια σύντομη παρουσίαση να σας κάνω. Την έχω κιόλας μοιράσει. Ονομάζομαι Πασκάλ Σάντα Κατερίνα. Είμαι Γενικό Διευθυντή τη ε, Oxfam ε, Magazin du Monde. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ για να σα παρουσιάσω την ε, οργάνωση μας και τι πιστεύουμε εμείς σε σχέση με την εμπορική πολιτική, τις εμπορικές πολιτικές. Είμαστε μια οργάνωση ισότιμου εμπορίου που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Βασίζεται στην γαλλόφωνη, δράζει μάλλον στο γαλλόφωνο Βέλγιο. Πρόκειται για εθελοντές που εργάζονται στα εμπορικά μας καταστήματα και είμαστε ένα δραστήριο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Δίκαιου Εμπορίου που συγκεντρώνει 400 οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς και του Γραφείου για το Δίκαιο Εμπόριο και είναι ένα, μια, ένας οργανισμός που αντιπροσωπεύεται σήμερα εδώ με τον Σέργη ε, Γοροπαλάν εδώ. Ε, το δίκαιο εμπόριο είναι καταρχάς ε, προϊόντα, ε, τρόφιμα, που προέρχονται από τον Νότο, διότι πρόκειται για εμπόριο με φτωχές χώρες ε, και ε, του Βορρά επίσης. Γιατί, γιατί στηρίζουμε την τοπική γεωργία και το γεγονός ότι η υδροθιωτική και παγκόσμια αλλαγή θα πρέπει να στηριχτεί από τα προϊόντα. Τα προϊόντα λοιπόν έχουν εμπορικό στόχο, ναι, ε, πρέπει να βοηθήσουν τους παραγωγούς να ζήσουν, αλλά έχουν και κοινωνικό ρόλο, δηλαδή να προωθούν αξίες. Εργαζόμαστε λοιπόν βασικά με μικρούς παραγωγούς, μικρής κλίμακας. Η Oxfam δηλαδή δεν εργάζεται, δεν συνεργάζεται άμεσα με τους γεωργούς, αλλά περνά από την Oxfam, Trade, από την Etikable. Και εδώ τονίζουμε το γεγονός ότι οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε γνωρίζουν τους ανθρώπους που φτιάχνουν το κάθε προϊόν. Δεύτερη πτυχή του δίκαιου εμπορίου είναι προϊόντα ε, βιοτεχνικά και εδώ εισάγουμε προϊόντα τα οποία προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο, από την Ινδία, από τη Σρι Λάγκα, όπως εδώ οι φωτογραφίες που βλέπετε. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει δίκαιο εμπόριο παρά μόνος για τα τρόφιμα, μιλάμε και για τις τράπεζες οι οποίες προσπαθούν να μπορευτούν δικαίως, αλλά όσο μας αφορά εμάς έχουμε να κάνουμε με την βιοτεχνία και ε, την χειροτεχνία. Ε, Υπάρχουν και, άλλες, ε, και άλλοι οργανισμοί όπως το Artisan du Monde, Solidar Monde στη Γαλλία. Ο οργανισμός μας υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Μιλάμε για μια πραγματική εμπειρία, για μια εμπορική δραστηριότητα διαφορετική που βασίζεται σε διαφορετικές αρχές. Οι αρχές αυτές φέρνουν ωφέλη γιατί μιλάμε για εμπόριο αλλά ε, δίνουν και ε, το μέσα διαβίωσης σε περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο που ασχολείται με την δίκαιη ε, γεωργία. Πρόκειται για ένα κίνημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλάμε για ένα μια πραγματική στήριξη, μια, ένα κίνημα πολιτών με ιδιαίτερη νομιμοποίηση στον χώρο του εμπορίου των προϊόντων. Συνεργαζόμαστε και ε, έχουμε 10 αρχές να δείτε ότι αυτές οι αρχές είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ε, παρατηρούμε ότι στηρίζοντας περιθωριοποιημένους παραγωγούς μειώνουμε την φτώχεια. Μία από τις αρχές είναι η ισότητα των φύλων. Η άλλη αρχή είναι η αξιοπρεπής εργασία. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτή η εμπειρία του δίκαιου εμπορίου ευθυγραμμίζεται με σημαντικό πλαίσιο που στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και από τους πολίτες όπως αυτό των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, Δεν είμαστε λοιπόν παρά ένας εμπορικός μόνο ένας εμπορικός οργανισμός, είμαστε ένας οργανισμός που θέλει να προωθήσει αξίες. Οπότε μέσα από το δίκαιο εμπόριο ε, δεν το, το, το βλέπουμε σε ένα στόχο για να στηρίξουμε μια εμπορική δραστηριότητα ε, για βιοτέχνες αλλά και γεωργού του Νότου, αλλά και ως ένα μέσο, βλέπουμε το εμπόριο, να καταγγείλουμε τις άδικες πρακτικές. Για παράδειγμα, δείξαμε, αποδείξαμε ότι υπάρχει συγκέντρωση εξουσίας στην ε, στον τομέα του χυμού πορτοκαλιού που προέρχεται, αποφύλεται μάλλον στις δασμολογικούς φραγμούς της ΣΥΠΑ και στην αγορά μας έχουμε ένα σωρό μάρκες από χυμούς πορτοκαλιού αλλά τρεις μόνο είναι οι μάρκες που εξάγουν από τη Βραζιλία τα πορτοκάλια. Ε, ε προτείνουμε λοιπόν ε, ε, προϊόντα από το δίκαιο, δίκαιη παραγωγή, δίκαιη ανάπτυξη και παρατηρούμε από την πηγή, την παραγωγή, την ε, κατανάλωση μέχρι και την ε, ρήψη των αποβλήτων. Υπάρχουν εναλλακτικέ και αυτέ θα πρέπει να στηρίξει ο περισσότερο κόσμο. Επίση, ε, κάνουμε ευαισθητοποίηση στους, για του πολίτε και μάλιστα για παράδειγμα με του προμηθευτέ έχουμε κάνει εκστατείε για την ισότητα των φύλων στην Ινδία και στο Μπαγκλαντέ, ενώ ταυτόχρονα έγιναν και εδώ στο Βέλγιο τέτοιε εκστατείε για την ισότητα των φύλων και έπειτα προσπαθούμε προσπαθούμε, αυτό που κάνω εγώ τώρα, να επηρεάσουμε τους υπεύθυνους για τη λήψη των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων. Έχουμε φυσικά ένα όραμα για ένα σύστημα που βασίζεται σε μια δημοκρατική κοινωνία και μια βιώσιμη οικονομία. Πιστεύουμε πως η φτώχεια βρίσκει την ρίζα της στις ανισότητες και ότι οι ανισότητες είναι καρπός πολιτικών επιλογών και οικονομικών αποφάσεων. Είναι ένα κακό νέο αυτό, αλλά και ταυτόχρονα και καλό νέο, γιατί εφόσον πρόκειται για επιλογή μπορούμε να προβούμε σε μια άλλη επιλογή. Το να έχουμε δηλαδή μια διαφορετική εμπορική πολιτική είναι δυνατόν, μπορούμε να δούμε ε, την πολιτική αυτή που είναι η πολιτική Trade for All της ε, κυρίας Επιτρόπου Μάλμστρομ είναι κάτι το οποίο ε, περιλαμβάνει ορισμένες θετικέ πτυχές γιατί υπάρχει και μία παράγραφος ολόκληρη για τα όσα αφορούν την βιωσιμότητα, την αναγνώριση της σημασίας μιας εμπορικής πολιτικής που βασίζεται σε αξίες, πράγμα που για μας είναι προφανές. Επίσης υπάρχει ένα τμήμα για την προώθηση του βιώσιμου δίκαιου εμπορίου που μάλιστα έγινε, έγινε και η δημιουργία ενός βραβείου για την, το ηθικό εμπόριο και αυτό στηρίζεται από τους πολίτες και ως κίνημα για το δίκαιο εμπόριο βρίσκουμε μάλλον συγγνώμη και μέτρα για, ε, ε, ε, για την αλυσίδα αξιών. Στηρίζουμε αυτή την, την παράγραφο. Ωστόσο, ε, λυπούμαστε γιατί τα περισσότερα αιτήματα που γίνονται προς τον ιδιωτικό τομέα βασίζονται πάντα σε μια εθελοντική προσέγγιση. Για μας αυτό δεν αρκεί. Γιατί η βελτιστοποίηση του ιδιωτικού συμφέροντος μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες, δηλαδή είναι ενάντια στο γενικό συμφέρον ε, μακροπρόθεσμα. Μπορεί δηλαδή να προχωρήσουμε από μια πλευρά γιατί θα κάνουμε επιλογή, θα επιλέξουμε τους στόχους μας ενδιαφέρουν, γιατί εδώ μπορεί κανείς να έχει βραχυπρόθεσμο κέρδος ε, και να αφήσουμε κατά μέρο αυτό που μας ενδιαφέρουν λιγότερο, γιατί εκεί η απόδοση του κεφαλαίου μας δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο θα θέλαμε. Για να μπορούμε όμως να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και παγκόσμια ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει μια πιο καθολική προσέγγιση ε, από όλους τους φορείς. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι για μας είναι σημαντικό το εμπόριο, ναι, αλλά με τρόπο που να είναι δίκαιο και να σέβεται τον άνθρωπο και τον πλανήτη πρώτα απ' όλα. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται πάντα. Γιατί πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Σήμερα άνθρωποι που ζουν σε ε, ειστερούσες περιοχές δεν έχουν τις συνθήκες για να βιώσουν σε βιώσιμο περιβάλλον λόγω μηχανισμών που δημιουργούν έλλειψη ισορροπίας και οδηγούν σε καταστάσεις τελείως άνησες, άδικες όπως άδικες τιμές και καταστάσεις αθέμητου ανταγωνισμού. Τελικά, μια ολόκληρη σειρά ανθρώπων, εργαζομένων, ε, ε, βιοτεχνών, γεωργών, ε, βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας παραγωγής και δουλεύουν υπό συνθήκε αναξιοπρεπή και συνθήκε διαβίωση αναξιοπρεπή και βρίσκονται κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Μάλιστα, πολλοί κόσμοι που παράγει την τροφή σε ολόκληρο τον πλανήτη υποφέρει από πείνα και οι έρευνε μα δείχνουν, είναι ετήσιε έρευνε που γίνονται από το 2010 και βλέπουμε σε αυτέ ότι 62 άνθρωποι οι πλουσιότεροι στον πλανήτη έχουν στην κατοχή του το ίδιο με το μισό των 3,5 δις των φτωχότερων στον πλανήτη. Δηλαδή 1% των πιο πλούσιων έχουν το ίδιο με το 99% υπόλοιπο της 100 του πλανήτη, κατοίκων του πλανήτη. Γι' αυτό λέμε trade for all. Ε, βέβαια, όλα αυτά δεν οφείλονται μόνο στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά το, οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να είναι ένα εργαλείο για την εξισορρόπηση αυτών των ανισοτήτων. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό οι εμπορικές συμφωνίες να σέβονται να δίνουν και να εγγυώνται το χώρο για τις ε, πολιτικές, ε, τις κοινοφελείς πολιτικές, ας πούμε η, πολιτική διατροφική, να ξέρουμε πώς παράγονται τα προϊόντα, ποια είναι η ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε, πολιτικές που επιτρέπουν να δημιουργηθεί και να προστατευτεί εργασία, ε, κλιματικές πολιτικές και βέβαια φορολογική πολιτική πιο δίκαιη. Θεωρούμε πως 7 σε 3 ε, δολάρια κρύβονται αυτή τη στιγμή σε παραδείσους φορολογικούς. Ένα τεράστιο κομμάτι φόρων λοιπόν που διαφεύγει από τα κράτη, που θα μπορούσαν με αυτά τα χρήματα να ασκήσουν προοδευτικές πολιτικές. Η νέα λοιπόν εμπορική πολιτική θα πρέπει να έχει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά όπως να προστατεύει τα εξαιρετικά καθεστώτα ή μέτρα ώστε να μπορούν λιγότερο προηγμένες χώρες να έχουν πρόσβαση στην αγορά και να μπορέσουν να καλύψουν την καθυστέρησή τους. Επίσης και είναι στόχος αυτού του πάνελ ότι πρέπει να συμφιλειωθεί ο πολίτης με τους δημόσιους θεσμούς και τους ιδιωτικούς θεσμούς, δηλαδή τις πολυεθνικές, καθιστώντας πιο διαφανείς τους μηχανισμούς ε, λήψης αποφάσεων, το είπα και πριν από λίγο, σε περίπτωση ρύθμισης ε, κάποιες διαφοράς, πιστεύουμε κυρίως στις χώρες μας ε, που έχουμε αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, ότι θα πρέπει να περνάμε από αυτό το σύστημα. Η ρύθμιση δηλαδή μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου, διαφοράς μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα θα πρέπει να γίνεται από τη δημόσια δικαιοσύνη. Και έπειτα, ε, για χρήματα που δεν κερδίζουμε, ποια είναι η επίπτωση στην ε, κοινωνία, στο περιβάλλον και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Για μας τελικά η απάντηση είναι σχετικά απλή. Εάν θέλουμε να έχουμε νομιμοποίηση, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε. Ε, και υπάρχουν πολλά πλαίσια που υπάρχουν. Υπάρχει COP21 που ε, ακόμα συζητείται και πάλι στο Μαρακέ, συμφωνίες για το κλίμα. Υπάρχει το πλαίσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια. Υπάρχει το πλαίσιο για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι εξαιρετικό πλαίσιο που μάλιστα ζητά την παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα για να συντονιστούν τα εμπορικά με τα αναπτυξιακά ζητήματα. Πράγμα το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στο εμπόριο. Ως ε, δίκαιο εμπόριο είμαστε βέβαια μέσα στα αγώνα στον ωκεανό, αλλά η μεγάλη μας περηφάνεια είναι ότι αποδεικνύουμε πως γίνεται να εμπορευτεί κανείς με τις αρχές του δίκαιου εμπορίου και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. κύριος Μπρέντιν τώρα. Μπρέντιν. Οικονομολόγος από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η ανάπτυξη του εμπορίου είναι το κλειδί για να βάλουμε τέλος στη φτώχεια. Πάντως αυτή η φράση θέλω να μας μιλήσετε. Βεβαίως, Πρόεδρε. Καταρχά, θέλω να συνεχίσω στα όσα είπε ο έρθω από το Ουσματικό Ταμείο για τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στο κοινοβουλευτικό δίκτυο και η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ για τη συζήτηση των θεμάτων που μα απασχολούν. Για να επανέλθω λοιπόν, η νομοποίηση του εμπορίου για την Παγκόσμια Τράπεζα απορρέει από τη σημασία του ως προς τον περιορισμό της φτώχειας. Είχαμε με τον ΠΟΕ συνέδριο για το ρόλο του εμπορίου στο τερματισμό της φτώχειας ακριβώς αυτό ήταν το θέμα και θα σταθώ σε αυτόν. Κοιτάξτε αυτή τη ε, φωτογραφία που σας δείχνω. Είναι τα σύνορα ανάμεσα στη Ρουάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Ε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα αυτά καθημερινά κυρίως γυναίκες και φτωχές γυναίκες. Ε, αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ταυτόχρονα υπάρχει και η πραγματικότητα που ζούμε στις ανεπτυσσεγμένες χώρες και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια σε αυτές χάρη στο εμπόριο. Δεύτερον, ε, βλέπετε μια γραμμή που ανεβαίνει, μια γραμμή που κατεβαίνει δεν ε, είναι διαφορετική η δική μου παρουσίαση από αυτές ε, που γενικά βλέπουμε σε οικονομικούς και εμπορικούς όρους. Ε, η πρώτη, το πρώτο διάγραμμα δείχνει την παγκοσμιοποίηση, παγκόσμιες εξαγωγές και ΑΕΠ που έχει αυξηθεί σημαντικά έως και τρίπλασια στην τελευταία 20 ετία, 20 ετία, 25 ετία και η μείωση της παγκόσμιας φτώχειας στη δεξιά στο δεξιά, δεξιο, δεξί διάγραμμα, που για μας σημαίνει πως το εμπόριο όσο αναπτύσσεται βοηθάει στη μείωση της φτώχειας, συμπιέζει τη φτώχεια στον κόσμο με την επόμενη διαφάνεια τα βλέπουμε νομίζω λίγο πιο ξεκάθαρα. Στο αριστερό κομμάτι της βλέπετε την Ανατολική Ασία και την Κίνα και τον περιορισμό του αριθμού των φτωχών στην Ανατολική Ασία που έχουν φτάσει μέχρι και να ε, έχει φτάσει μέχρι και να εκμηδενιστεί. Ένα, τρισεκατο... δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν φτάσει να βγουν από τη φτώχεια στην τελευταία 20 ετία. Στη δεξιά όμως, ε, στο δεξί μέρος της διαφάνειας βλέπετε την πρόκληση που παραμένει ακόμη ενώπιόν μας, αυτούς που ζουν σε ακραία φτώχεια. Πάλι η Ανατολική Ασία, αν και μέχρι το 2030 θα έχουν ξεφύγει από τη φτώχεια σε μεγάλο βαθμό. Για το 2030 η ακραία φτώχεια θα αφορά μόνο την Αφρική, από ό,τι λένε οι προβλέψεις μας. Και θα είναι τραγωδία αυτή τη στιγμή το να παρεμποδίσουμε ε, τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν για να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση τώρα. Πώς δηλαδή μπορούμε να επιτρέψουμε στην παγκοσμιοποίηση να θέσει ένα τέρμα στην ακραία φτώχεια στις περιοχές όπου αυτή παραμένει υπαρκτή. Η Αφρική αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση γιατί έχει αυξηθεί σημαντικά το εμπόριο την τελευταία δεκαετία εκεί, χωρίς όμως να φέρει η αδίποτε εξέλιξη, πολύ περιορισμένε πάντως, σε σχέση με τη φτώχεια, με το, με το επίπεδο της φτώχειας. Είναι λοιπόν το κλειδί μεν, αλλά όχι η εγγύηση για το τέλος της φτώχειας. Και έτσι περνώ στην επόμενη διαφάνεια, για να αναπτύξω τώρα αυτή τη θέση. Το εμπόριο λοιπόν το συζητούμε και σκεφτόμαστε συνήθως ότι αποτελεί ένα παράγοντα υποστήριξης της ανάπτυξης, αλλά μπορεί να έχει κεντρική σημασία για τον περιορισμό της φτώχειας και σε άλλους όρους. Ενίσχυση της θέσης των γυναικών και χειραφέτηση αυτών. Εκατοντάδες χιλιάδων γυναικών έχουν βρει ε, απασχόληση και θέση στη ζωή ε, ε, ειρήνη και σταθερότητα. Ρουάντα θα σας πω ως ε, σύνθημα. Η αστάθεια και οι συγκρούσεις ενισχύουν τη φτώχεια, περιορίζουν το ΑΕΠ. 90-95% των φτωχών του κόσμου του 2030, το 2030 θα ζουν σε ασταθή κράτη. Αν λοιπόν δεν προχωρήσουμε ε, χάρη στο εμπόριο στη σταθερότητα, ή μάλλον το εμπόριο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση σταθερότητα, θα έχουμε ακόμη πολλού φτωχού. Με πολλού τρόπου λοιπόν μπορεί να επηρεάσει τη φτώχεια, όπω είπα, χειραφέτηση, ασφάλεια διατροφική, ειρήνη, σταθερότητα κτλ. Όλα αυτά μπορούν να ε, σε όλα αυτά μπορεί να συμβάλλει το εμπόριο. Είναι ένα κλειδί λοιπόν, ένα κλειδί που μπορεί να ανοίξει πόρτες αλλά δεν αρκεί μόνο του και αυτό μας το έχει αποδείξει και η εμπειρία από την Αφρική τα τελευταία 15-20 χρόνια με την ε, ιδιαίτερα σημαντική θέση που έχουν στο εμπόριο των Αφρικανικών κρατών τα ορυκτά τα τελευταία χρόνια. Και περνώ στην επόμενη διαφάνεια για να σας παρουσιάσω τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί και έτσι δεν είναι σε θέση να ωφεληθούν από το εμπόριο, από τις εμπορικές συναλλαγές, κάτι το οποίο πρέπει αντίστροφα εμάς στις πλούσιες χώρες να μας ε, προβληματίσει ως προς τα ωφέλη που έχουμε από την παγκοσμιοποίηση και την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων. Προς, πρέπει λοιπόν να δούμε το, την αντίστροφη εικόνα. Ποιος είναι αυτός που ωφελείται από την παγκοσμιοποίηση και την ενίσχυση του εμπορίου ή ποιο είναι αυτό ο οποίο στερείται τα ωφέλη ε, της, ε, του εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης. Τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία περιορίζουν τον φτωχό. Ο φτωχός καταρχάς ζει στην Ήπεθρο, επομένως είναι αποκομμένος από του συνήθεις δρόμους του εμπορίου, πρώτο χαρακτηριστικό. Δεύτερον, επί το πλήστον εργάζεται και διαβιώνει σε άτυπες συνθήκες Επομένως δεν μπορεί να ωφεληθεί από τα επίσημα κανάλια ε, του εμπορίου. Επίσης, όπως είπα, οι περισσότεροι φτωχοί ζουν σε ευάλωτα και ασταθή κράτη με συγκρούσεις και αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν τη φτώχεια τους. Και τέταρτο, η ανισότητα ως προς το φύλλο. Πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες ζουν στη φτώχεια, χάρη στο εμπόριο μπορούν να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση εμπλεκόμενες σε εμπορικές δραστηριότητες. Για την Παγκόσμια Τράπεζα λοιπόν αυτές τις προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε απάντηση στην ακραία φτώχεια έως το 2030, για να έχουμε θέσει ένα τέρμα στην ακραία φτώχεια στο 2030, που είναι ο στόχος μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν συγκεκριμένα στην επόμενη διαφάνεια. Πρέπει να περιοριστεί το κόστος του εμπορίου μεταξύ των κρατών, δασμοί και μη δασμολογικά εμπόδια σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριμένες περιφέρειες ε, Ασία, νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας και το καθεξής, αλλά και ανεπτυγμένες χώρες που μπορούν να μειώσουν το κόστος που προξενείται από τις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης στο ιστορικό των κρατών Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα προς τον περιορισμό της φτώχειας, πρόσβαση σε αγορές, συνδεσιμότητα, εξυγχρονισμός. Ε, Επίση, πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και να περιορίσουμε του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί και δεν πρέπει να του παραγνωρίσουμε. Είναι τεράστιοι οι κίνδυνοι που και έτσι δεν μπορούν οι φτωχοί να ε, ωφεληθούν από το εμπόριο. Ένας ε, γεωργό, σε παραδείγμα, τη μικρή γεωργική εκμετάλλευση που απλώ παράγει τα το ζήν μπορεί να έχει κάποια ωφέλη από, την, ε, από τις συναλλαγές σε μια συγκεκριμένη συγκομιδή, σε ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, αλλά ε, η αστάθεια καιρική ή ε, κάποια κακή συγκομιδή σε συγκεκριμένη χρονιά τον φέρνει στο χείλος της ακραίας φτώχειας. Και άρα χρειάζεται να κοιτάξουμε ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι για να μπορέσει ο καθένας να προχωρήσει φερρυπίν στην εξειδίκευση και στην παραγωγή ενός μόνο προϊόντος χωρίς να φοβάται ότι θα εκτεθεί στους κινδύνους αυτούς. Επίσης το περιβάλλον, η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη συμμετοχή στις εμπορικές συναλλαγές. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η Ρουάντα έχει επενδύσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Ένα εκατομμύριο παιδιά στη Ρουάντα τώρα έχουν φτάσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακόμα και στην τριτοβάθμια. Τεράστια επένδυση. 60.000 θέσει εργασία θα χρειαστεί όμω η Ρουάντα όταν έρθει η ώρα αυτά τα παιδιά να τελειώσουν τι σπουδέ του και να αρχίσουν να δουλεύουν. Πού θα τι βρουν τι θέσει εργασία τα παιδιά αυτά. Το εμπόριο λοιπόν θα έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Βεβαίω η μετανάστευση πρέπει να το δούμε και αυτό και ξέρω ότι δεν, δεν εξετάστηκε αρκετά το θέμα της μετανάστευσης αλλά είναι δίδυμη αδελφή θα έλεγα του εμπορίου. Ε, εάν λοιπόν ε, βλέπουμε μια πολύ καλή επιλογή που είναι η επένδυση στην εκπαίδευση ε, πώς θα βρεθεί δουλειά για τους ανθρώπους αυτούς. Και εκεί το εμπόριο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και εν τέλει χρειάζονται καλύτερα δεδομένα για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις συνέπειες του εμπορίου. Όταν κανείς βρίσκεται στην Ήπεθρο, δρά μόνο σε άτυπο, στην άτυπη οικονομία, δεν μπορεί να ωφεληθεί από το εμπόριο. Άρα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και μπορούμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα και χάρη στην νέα τεχνολογία, τα νέα μέσα, τους δορυφόρου, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να παρακολουθούν πολύ καλύτερα δηλαδή τις συνέπειες επί παραδείγματι των οικονομικών εταιρικών σχέσεων στην φτώχεια για να κάνουμε και σχετικές προσαρμογές και για να ξαναγυρίσω στην αρχική μου φωτογραφία μια εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε ως φαινόμενο εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακραία φτώχεια σε περιοχές όπως είναι η Ρουάντα, όπως είναι η Ουγγάντα, όπως είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εάν δεν αλλάξουμε τις επιλογές αυτοί οι άνθρωποι θα υποφέρουν. Τι μπορούμε να κάνουμε σχέση με τα σύνορα αυτά και να βελτιώσουμε τι επενδύσει γιατί οι, οι, οι υποδομές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ε, για να καταλάβετε επαρκή υπόστεγα που να προστατεύουν τα προϊόντα. Θέλει κανείς να κάνει συναλλαγές σε στάρι, ε, εάν δεν έχει κατάλληλα υπόστεγα την ώρα που θα πιάσει η βροχή, το στάρι που θα καταστραφεί. Δεν υπάρχουν υποδομές σε τουαλέτες, δεν υπάρχουν υποδομές σε δρόμους. Απλά πράγματα. Πρέπει οι κανόνες επίση και οι διαδικασίε να απλουστευτούν, να γίνουν πιο διαφανείς, να ανοίξουν οι ευκαιρίε και να κλείσει οποιαδήποτε ευκαιρία είτε εκβιασμού είτε δωροδοκίας και βεβαίως να επιτραπεί λειτουργία χωρίς ε, προσκόμματα, χωρίς εμπόδια των οργανισμών που δρούν διασυνοριακά. Νωρίτερα εξετάθηκε περισσότερο το θέμα της δωροδοκίας και της διαφθοράς, μα ακριβώς εδώ πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις, στα σύνορα δηλαδή. Αν δεν δώσουμε στα σύνορα ε, λύσεις οι οποίες θα αποδιαρθρώσουν την διαφθορά και τη δωροδοκία δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτά είναι τα κύρια μελήματα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αυτά είναι η αυτοί είναι κύριοι για την ανάπτυξη ενός εμπορίου το οποίο θα θέσει τέρμα στην ακραία φτώχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Λάγκε. Και πριν παραχωρήσω το μικρόφωνο. Στους συναδέλφους να πρέπει να σας πω ότι έχω κάπως μπερδευτεί. Γιατί από τη μια πλευρά φαίνεται ότι είναι λογικό, δεν μπορούμε να κλείσουμε τις αγορές μας, υπάρχει παγκοσμιοποίηση και αυτό κατέστη σαφές από όλους. Α, είναι μια αυταπάτη το να λέμε ότι θα κλείσουμε τις αγορές. Το εμπόριο είναι απαραίτητο, όμως τώρα άκουσα από σχεδόν όλους ότι το εμπόριο λειτουργεί μόνο υπό όρους παιδεία, κατανομή των ωφελών, η εμπορική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεπής με τις άλλες μας πολιτικές. Ε, αναφέρθηκε και το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Η ερώτησή μου είναι τι γίνεται ε, αν δεν πληρώνται οι όροι. Τι θα κάνουμε, αφήσουμε τον πόριο στην άκρη, μόνο του, στην ησυχία του. Αυτό δεν γίνεται. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους εταίρους ώστε να φτιάξουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος να ωφεληθεί από το εμπόριο. Μια μικρή ερώτηση αλλά και μεγάλη ερώτηση προς όλους. Ο κύριος Φιέλνερ και μετά η Μαρία Ρένα. Σαφώ η ευρωπαϊκή ε, εμπορική πολιτική, η χάραξη πολιτικής είναι, διανύει μια υπαρξιακή κρίση. Πάντω δεν ακούω να λέτε περισσότερο προστατευτισμός. Θέλετε όμως να προστατεύσετε όμως από καιρού ει καιρού και εδώ ε, τους εμπόρους. Αυτό στο οποίο εγώ είμαι αντίθετος είναι αυτή η έννοια που πολύ συχνά λέμε ότι πρόκειται για νέο φαινόμενο ότι είναι κάτι που ξαφνικά προέκυψε. Όχι, λυπάμαι. Ε, Φρέντρικ Μπαστιάτ, Manchester Liberals, εκεί, αυτοί ήταν ε, οι αγώνες που είχαν ε, στις, στο κοινοβούλιο τους και ακριβώς αν διαβάσετε τις συνομιλίες, ακριβώς για την κατανομή του πλούτου ήταν η, η συζήτηση. Και ναι, μπορούμε να ψηφίσουμε για την εμπορική πολιτική, αλλά όχι για όλα τα όλα. Αλλά ακόμα και η αντιπολίτευση υπήρχε. Η, Επαναλαμβάνεται η ιστορία και κέρδισαν και ε, καρπώνονται τα ωφέλη. Και ποιο σήμερα θα έλεγε ότι μακάρι να ήμουν στην πλευρά των χαμένων. Αλλά ξαφνικά ο κόσμος όλα θα τα ξεχνάει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν είμαστε στον 14ο αιώνα. Το περάσαμε αυτό. Και ο κύριε Ρέιτερ είπατε πολλά σωστά για την πολιτική ανταγωνισμού, για την κοινωνική πολιτική, αλλά ας πούμε η βοήθεια για την προσαρμογή στο εμπόριο ή το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο επικρίναμε στο πλαίσιο του ΗΠΑ, είναι ακριβώς αυτή η βοήθεια για την προσαρμογή στο εμπόριο. Δηλαδή δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που ήταν μέσα στο πρόγραμμα και αυτούς που δεν ήταν. Αλλά μπορεί αυτό να είναι το πρόβλημα των ομοσπονδιακών προγραμμάτων. Και ε, επίσης πιστεύω πως και εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί σημαίνει ότι το εμπόριο είναι το πρόβλημα. Ποιος θα σκεφτόταν να πούμε πρόγραμμα προσαρμογής για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιγράφουμε τα πράγματα με τρόπο ε, ώστε τελικά ο κόσμος να πιστεύει πως το εμπόριο είναι το πρόβλημα. Και στρέφουμε στην τελευταία μας ομιλητή. Για να καταλάβω, αν ακούσω αυτό που λέτε, εσείς περιγράφετε, λέτε ότι ο κόσμος υποφέρει ο κόσμος δεν υποφέρει μάλλον από την παγκοσμιοποίηση, αλλά ότι επειδή δεν είναι κομμάτι της παγκοσμιοποίησης. Γιατί πολλοί λένε από αυτό το επιχείρημα, ναι, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι το εμπόριο είναι κακό ή η παγκοσμιοποίηση είναι κακή. Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μέρος τη παγκοσμιοποίηση και εξακολουθούν να υποφέρουν όπως και πριν την παγκοσμιοποίηση και θα συνεχίσουν για πάντα να υποφέρουν εάν δεν ε, το επιδιώξουμε. Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις διάφορες παρεμβάσεις. Ε, εγώ ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω πως εδώ υπάρχει έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά του εμπορίου. Θα ήταν παράλογο ως Ευρωπαίος να είναι κανείς αντίθετος στο εμπόριο. Είμαστε η πρώτη οικονομία που ζει από τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Θα ήταν λαϊκιστικό να πούμε ότι αντιτιθέμεθα στο εμπόριο. Αυτό είναι μια πρώτη, μια πρώτη παρατήρηση, γιατί είναι σωστό να διορθώνουμε, γιατί έχουμε κάποιες φορές την εντύπωση πως επικρατούν παρεξηγήσει σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκουμε. Όμως θα μπορούσαμε αντίθετα να είμαστε υπέρ του εμπορίου, αλλά να έχουμε να διατυπώσουμε επικρίσεις σε σχέση με τις εμπορικές πολιτικέ διότι οι εμπορικέ πολιτικέ μπορεί να δημιουργήσουν μια επιτάχυνση, να προκαλέσουν μια επιτάχυνση φαινομένων που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Δηλαδή τα φαινόμενα ανισότητα που ζούμε σήμερα μαζικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκόσμια. Το θέμα λοιπόν είναι οι εμπορικέ μα πολιτικέ οι σημερινέ, όχι οι χθεσινές, οι σημερινέ, ανταποκρίνονται στους στόχους που που πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε σήμερα. Ναι, η σημερινή κατάσταση δεν είναι η ίδια με τη μεταπολεμική. Βρισκόμαστε σε νέες καταστάσεις, νέες τεχνολογίες, σε παγκοσμιοποίηση πολύ πιο γρήγορη. Οι δικέ μα εμπορικές πολιτικές λοιπόν ανταποκρίνονται στους στόχου και στις προκλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να, να, να θέσουμε το ερώτημα έτσι. Ένα άλλο που, για το οποίο συμφωνώ είναι ότι οι εμπορικές πολιτικές δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα, προφανώς. Το μόνο ζήτημα είναι πως έχουμε εδώ την εντύπωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι προχωράμε κουτσά. Δηλαδή βασιζόμαστε ε, στις εμπορικές πολιτικές που δεν είναι αναγκαστικά προσαρμοσμένες στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί είναι η μόνη πολιτική επί τη οποία μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση και να έχουμε και μια πλειοψηφία ενώ αντίθετα για όλα τα άλλα για την οργάνωση της αλληλεγγύης, των επενδύσεων, της βιομηχανικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν καταφέρνουμε να έχουμε συνένεση. Αυτό είναι που μας δημιουργεί τις δυσκολίες. Η ισορροπία ανάμεσα σε μια πραγματική οικονομική και εμπορική πολιτική που θα έπρεπε να έχουμε και τις υπόλοιπες πολιτικές της ευημερία που πρέπει να εγγυηθούμε στην Ευρώπη αλλά και, συμφωνώ μαζί σας, στον υπόλοιπο κόσμο και στην Αφρική μεταξύ άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρω ότι είμαστε στην Ίντα και ότι ασχολούμαστε με την εμπορική πολιτική, αλλά πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας και να πούμε ότι πρέπει να συντονιστούν και άλλε πολιτικές. Ευχαριστώ. Σόλτ. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. για το παράδειγμα που δώσατε για την διαπραγματευτική εντολή. Πώς μεταφράζουμε την ζήτηση αυτή, τις προτάσεις αυτές, τις εναλλακτικές αυτές επιλογές, δεδομένου του πλαισίου όπου το εμπόριο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, μεγάλες επιχείρησεις όπως η Apple ή άλλοι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι συμφωνούν με τις αρχές που, βάζουν αυτή, που βάζει αυτή η ζήτηση. Δηλαδή πώς θα επανοργανώσουμε αυτό το διεθνές πλαίσιο. Ευχαριστώ την Αράντσα Σάντσες. Η απέτησή σας ότι το εμπόριο πρέπει πάντοτε να είναι ανοιχτό, inclusive, δηλαδή τι σημαίνει αυτό όμως. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα σύνολο κανόνων προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν αναφέρομαι στην σημερινή Ευρώπη, αλλά περισσότερο στους εμπορικούς μας εταίρους. Ελέγχθη προηγουμένως ότι χρειάζεται πρόσβαση στην τεχνολογία και ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του ενισχυμένου εμπορίου. Εγώ έχω ορισμένα αντεπιχειρήματα. Παράδειγμα, στην εποχή που αναπτύσσονταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ βρισκόμουν στην Ιαπωνία και εκεί ήταν απολύτως κλειστή η κοινωνία εκεί. Δεν μπορούσε να εισαχθεί υπολογιστής από την αλλοδαπή. Οι δε ιαπωνικοί υπολογιστές ήταν άχρηστοι. Αυτός ο απομονωτισμός οδήγησε τελικώς όμως την Ιαπωνία να αχθεί στο υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας που βρίσκεται σήμερα. Τώρα, άλλο παράδειγμα. Γερμανία μετά τον πόλεμο. Δεν είχαμε εμπορικές συμφωνίες τότε από, το, τον δικό μου τομέα, δηλαδή την ε, οργάνωση δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο να επιτευχθεί δηλαδή ο ρόλος που έπαιξε η Γερμανία τη δεκαετία του 90 και μετά, εάν υπήρχαν τότε τέτοιες συμφωνίες, διότι η αγορά, όχι νομοθετικά, αλλά ουσιαστικά ήταν απομονωμένη. Τα φέρνω αυτά ως παραδείγματα, διότι θέλω να εξηγήσω ότι καμιά φορά για να μπορέσει να πάρει μπρος μια βιομηχανία, χρειάζεται μια προστατευμένη αγορά, ώστε να μπορέσει να συλλεχθεί το αναγκαίο κεφάλαιο, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια τέτοια βιομηχανία. Ζητώ, παρακαλώ να το λάβετε υπόψη αυτό. Το άνοιγμα των αγορών, ιδίω για αναπτυσσόμενε ή χώρε κατοφλίου, μπορεί να οδηγήσει και σε σε αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Και Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε η Μαρή Αρενά. Νομίζω ότι πολλοί που λένε ότι είναι αντίθετοι με το εμπόριο, στην πραγματικότητα είναι αντίθετοι με τις εμπορικές πολιτικές. Διαφορετικά πράγματα. Μιλώ από την εμπειρία μου σχετικά με την Βρετανική έξοδο και με το τι έγινε χθες στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, η δική μου εκλογική περιφέρεια θα μπορούσε να συγκριθεί με την Πενσιλβανία. Έχουμε δηλαδή ε, εξαγωγικό πλεόνασμα. Είμαστε η μοναδική αγγλική περιφέρεια η οποία εξάγει περισσότερα από όσα εισάγει. Και όμως είχαμε τις περισσότερες ψήφους υπέρ της εξόδου leave votes, να φύγουμε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματα τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που βλέπουμε τώρα στις ΗΠΑ. Έχουμε λοιπόν αυτό το παράδοξο που παραλύει το διεθνές σύστημα και ενδεχομένως θα παραλύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα δηλαδή στην ανάγκη επαναρρύθμισης της οικονομίας μας και στην έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού σχετικά με την νέα αυτή ρύθμιση στο διεθνές επίπεδο. Έχει τόσο αποκλίνει η οικονομία μας πέρα από τα ρυθμιστικά πλαίσια που έχει αποσυνδεθεί πλήρως. Με εξέπληξαν οι παρουσιάσεις σας που μου φάνηκαν όλες να αναφέρονται στην σημασία του εμπορίου. Δεν αναφέρθηκαν όμως το πώς θα αποκαταστήσουμε την νομιμοποίηση του εμπορίου και πώς θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και των ανθρώπων της εκλογικής μου περιφέρειας στην βορειοανατολική Αγγλία ή των ανθρώπων που ζουν στην Πενσιλβάνια ή άλλων κοινοτήτων που θεωρούν ότι δεν έχουν απολαύσει ωφέλη ισοτήμως από την παγκοσμιοποίηση. Και η ανισότητα αυτή είναι ε, το κλειδί για να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αρχίσει καν το ρολόι, έτσι, το χρονόμετρο δηλαδή, να μετά το χρόνο μου. Ε, πάντως, ένα θέμα ακόμη. Η εμπειρία της Ένωσης δείχνει ότι η αδυναμία της κοινωνικής διάστασης είναι το κλειδί. Εξεπλάγει με αυτό που είπε ο κύριος Ράιτερ, ότι δεν είμαστε ιεραπόστολοι της νομοθετικής ρύθμισης και σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα. Πώς όμως θα εξορροπήσουμε το γεγονός ότι όλοι έχουμε αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο ε, την δέσμευση να ε, υποστηρίξουμε τους στόχους της βιωσιμότητας τους στόχους ε, της Συμφωνίας του Παρισιού, όμως τα υπόλοιπα είναι όλα οικειοθελή. Εκεί είναι η δυσκολία. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, ιδίως σχετικά με τα όσα είπαμε για την εναλλακτική εμπορική εντολή. Εγώ δεν το πιστεύω, ναι. Τέλος, είμαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις ε, παρεμβάσεις τους. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιο βαθμό όπως ε, μιλάμε για μια εμπορική πολιτική για όλους, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και μια οικονομική πολιτική για όλους. Γιατί αν δεν πάνε χέρι-χέρι και αν δεν ξεκινήσουμε από αυτή την αρχή πώς, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη που θα προσφέρει ε, ε, δυνατότητες και ευκαιρίες, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που να έχει σκεφτεί την συσχέτιση μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής ε, ώστε να επιτυχθεί πραγματικά μια παγκοσμιοποίηση για όλους γιατί κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι αυτό που τονίζει η παγκοσμιοποίηση είναι οι δυνατότητες ε, και οι δυνάμεις των διαφόρων ομάδων της κοινωνίας και γι' αυτό η εμπορική πολιτική είναι αυτή το, η αιχμή του δώρατος της οποίας συγκεντρώνονται όλες οι επικρίσεις κατά της παγκοσμιοποίησης. Ίσως λοιπόν επειδή υπάρχει έλλειψη ε, ε, δεξιοτήτων ε, αλλά και δυνατοτήτων ε, στην, σε κρατικές δομές για να μπορέσουν δηλαδή με τις εκπαιδευτικές τους πολιτικές ή τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές για την κοινοτομία να καλύψουν την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί. Εάν δεν υπάρξει συντονισμός λοιπόν ανάμεσα σε όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και τον φόβο των πολιτών που, ότι θα χάσουν ε, τις ε, συνθήκες διαβίωσής τους, ε, οι οποίες θα επιδεινωθούν αν δεν... Είναι δυνατόν, υπάρχει κάποιος τέτοιος οργανισμός. Το έχει σκεφτεί αυτό. Ευχαριστώ. Μια ακόμη ερώτηση από δικής μου πλευράς. Το κίνημα για το δίκαιο εμπόριο και το παραδοσιακό εμπόριο φαίνεται να προχωρούν σε δύο παράλληλους δρόμους. Δεν θα ήταν καλύτερο να τα ενώσουμε, έτσι ώστε το δίκαιο εμπόριο να ήταν όλο και πιο τακτικά κομμάτι του συμβατικού εμπορίου. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και άλλη μια ερώτηση από τον τοίχο του Twitter. Η μία μάλιστα σχετίζεται με την ερώτηση της κυρίας Ντάρλινγκ. Πιστεύετε ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα οι όροι που προβλέπονται στις εμπορικές συναλλαγές και δεύτερον τι είδους ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που θέλουν να επενδύσουν στην αηφορία. Ο κύριος Ράιτερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολλές οι ερωτήσεις ε, και πολύ συγκεκριμένες. Πολλές από αυτές. Πέντε λεπτά μου δίνετε. Λοιπόν, για να κερδίσω χρόνο, ξεκινώ με την ερώτηση της ε, κυρίας Ντάρλινγκ. Ακριβώς ε, εδώ ήθελα να εστιάσω την διαφοροποίηση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πολιτικής για το εμπόριο. Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε και πολλά απορρέουν από την ανεπαρκή απάντηση στο φόβο, στις ανησυχίες, στα μελήματα ε, εύστοχα για τις ε, αδικίες. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο. Τώρα τυχαίνει να μιλάμε για το εμπόριο, αλλά και η αυτοματοποίηση μπορεί να φέρει τα ίδια, ε, τις ίδιες συνέπειες. Η εισαγωγή της μηχανογράφησης που θα εξαφανίσει τόσες θέσεις εργασίας Πρέπει να κάνει κανείς κάτι, διαφορετικά θα το βρει μπροστά του στις προσεχείς εκλογές. Επομένως, πολλά είναι, πολλοί είναι τομείς δραστηριότητα και πολιτικής. Δεν είναι μόνο ε, το εμπόριο μια ευκαιρία για την κοινωνία, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίσουμε ότι είναι ένα διαναμετικό και μπορεί να φέρει ισότητα, περισσότερη ισότητα, ιδιαίτερα εάν προχωρήσει μέσα από κατάλληλες πολιτικές εθνικές. ένα παράδειγμα. Δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτή η πρακτική που είναι τόσο κοινή στις ανεπτυγμένε χώρες, όπου είναι πολύ με, λίγες οι μεγάλες επιχειρήσεις με δυνατότητα και δυναμικό κινητικότητα και άρα και απορρόφηση των πόρων, οι οποίες ωφελούνται αλλά δεν μπορεί να ωφεληθεί κανεί άλλος. σε αυτό δεν πρέπει να δοθούν απαντήσει. Και επίση η αρχική και η γενική ερώτηση του κύριου Λάγκε να μην κλείνουν οι αγορές αλλά να κινούμεθα αν είναι κατάλληλε οι συνθήκες. Δεν νομίζω ότι είπε κανεί κάτι τέτοιο. Το εμπόριο φέρνει, νομίζω ότι όλοι αυτό είπανε, φέρνει καλά αποτελέσματα. Αλλά αν θέλουμε να είναι και πολιτικά βιώσιμα αυτά και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα ωφελούνται, όχι οι λίγοι, ούτε καν οι πολλοί ει βάρος των λίγων αλλά ότι θα ωφελούνται όλοι από το εμπόριο, τότε χρειάζονται ακόμη περισσότερα μέτρα στήριξη και πολιτική. Έχει φέρει αποτελέσματα το εμπόριο, το έχουν πει πολλοί από του ομιλητέ μα. Να σα δώσω ένα ακόμα στοιχείο. 62% τη αγοραστική αξία του φτωχού Αμερικανού εξαρτάται από το ελεύθερο εμπόριο. Το 62%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αδίποτε πρόταση για ε, εισαγωγή τελωνιακών δασμών θα είναι η πιο οπισθοδρομική φορολογική πρόταση, η δασμολογική πρόταση που θα μπορούσε κανείς ποτέ να διανοηθεί, εάν εισαχθεί κάτι τέτοιο τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε απαντήσεις από το γεγονός ότι πολλές φορές λίγοι ή και πολλοί πλήττονται από τα μέτρα αυτά. Για τον κύριο Φιέλνερ, να έχετε δίκιο, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα σε μια συζήτηση πολιτική, υπεύθυνη και αποτελεσματική. Εδώ έχουν ευθύνη οι πολιτικοί να δώσουν ε, τον, ε, το ρυθμό θα έλεγα να δώσουν τις απαντήσεις. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τόσο κρίσιμες ε, εκλογές στη Σουηδία συχνά, αλλά είχαμε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση το 1989 και αφορούσε τους θελωνιακούς δασμούς και την κατάργησή τους. Άρα καλούνται οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή Τη ιστορία του να δώσουν απαντήσει κρίσιμε. Επικαιροποίηση τη πολιτική για το εμπόριο. Φυσικά, το status quo ούτω ή άλλω αποτελεί οπισθοδρόμηση και για την πολιτική εμπορίου και πρέπει να δώσουμε απαντήσει. Πρώτα απ' όλα με βάση τις προτιμήσεις των πολιτών μας, αλλά και σε δεύτερο βαθμό στις εξελισσόμενες συνθήκες του εμπορίου. Πρέπει διαρκώς να επικαιροποιούμε λοιπόν και να κάνουμε κάτι καλύτερο κάθε φορά. Ένα πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα είναι το πώς θα εξισορροπηθεί η κοινωνική διάσταση με την αηφόρο ανάπτυξη. Θα σας πω το εξιστό εμπόριο και το ανοιχτό εμπόριο είναι ενσωματωμένο, είναι ε, όρος εκτρώνου κάνευ και συστατικό στοιχείο του, της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτό το συμφωνήσανε και με τους στόχους του 17 οι ηγέτες πέρυσι δεν υπάρχει σε αυτό αμφισβήτηση. Μπορεί να μην το βλέπουμε σε όρους ε, εκλογικών αναμετρήσεων αυτή την βεβαίωση, αλλά οι πολιτικές οδηγίες, πολιτικές ε, κατευθύνσεις έχουν ήδη δοθεί από τους ηγέτες. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα να εξορροπήσουμε σε σχέση με συγκεκριμένες απαιτήσει για ορισμένε χώρε. το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να μεριμνείτε ιδιαίτερα για αυτό που επισημαίνουν τα αναπτυσσόμενα τα κράτη ιδιαίτερα Οι φυστάμενε συμβάσει. Είμαι υποχρεωμένο, καθώ ομιλώ εκ μέρου των ΗΠΑ, να το επισημάνω αυτό, αλλά και το Συμβούλιο των ΗΠΑ για το δικαίωμα τη ανάπτυξη και εσείς το κοινοβούλιο σας λέει ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της ρύθμισης. Ναι, όπως και τα αναπτυσσόμενα κράτη όμως, τα οποία μπορεί να μην έχουν το δικαίωμα να κάνουν dumping ή να παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες, αλλά έχουν το δικαίωμα να εισάγουν ειδικού τους κανόνες. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε τόσο τον ιεροκήρυκα, γιατί εν τέλει ο μόνος τρόπος να λειτουργήσουν αυτές οι κοινωνίες, όλες οι κοινωνίες καλά στον σημερινό κόσμο, είναι να συνεργάζονται. Και αυτό σημαίνει ταπεινότητα και σημαίνει εφουγκράζω με τον άλλον πριν ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τα, αναπτυσσόμενα, τα ανεπτυγμένα κράτη να εκφράζουν όλο και περισσότερε απαιτήσει σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε υπάρχει λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια υστερόβουλη ε, πρόθεση από τα ανεπτυγμένα κράτη να καθυστερήσουν την ανάπτυξη των αναπτυσσομένων κρατών. Τουλάχιστον αυτά έτσι αισθάνονται, ότι κάποιο προσπαθεί να παρεμποδίζει την προοδό του για να τα εκμεταλλεύεται ακόμη περισσότερο. Και αυτό μπορείτε να το κερδίσετε μόνο και να πείσετε μόνο, εάν αντί να του κάνετε το κήρυγμα, συνεργαστείτε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο. Ε, κυρία Κονσάλε. Δύο βασικέ αλλαγέ βλέπω σε σχέση με τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μπαστιά και και την περίοδο στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα και την κατάσταση που παρουσίαζε η Γαλλία. Μια, διαφορά ήταν η διασύνδεση των οικονομιών που είναι διαφορετική σήμερα από ό,τι ήταν κάποτε στο παρελθόν. Τότε μιλούσαν για κεριά και για ε, δημητριακά. Τώρα όμως μιλούμε για αντανακτικά των iPad και αυτό, αυτή η διαλειτουργικότητα είναι που πρέπει να μας απασχολήσει και την κατανοήσουμε σωστά. Εάν θέλουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ίδια αυτά επιχειρήματα τα οποία έχουν σχέση και με τις αλλαγές στους οικονομικούς και κοινωνικούς ιστούς που προέρχονται από την οικονομική πρόοδο και το άνοιγμα. Η δεύτερη θεμελιώδης διαφορά και αυτή είναι που με ανησυχεί είναι όταν ακούω όταν ζούμε, ότι ζούμε τώρα σε μια post-factual κοινωνία, διότι τελικώ η οικονομία ε, έχει σχέση με τα facts, με τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομία με tweet. Χρειάζεται να εξηγήσουμε, να δώσουμε γεγονότα, ε, αριθμού. Αυτό είναι ο παιδαγωγικό ρόλο τη οικονομία. Για να εξηγήσουμε λοιπόν στους πολίτες, ξεκινώντας από τα βασικά της πολιτικής, να εξηγήσουμε στον πολίτη τι λειτουργεί και αποδίδει, τι δεν αποδίδει και δεν λειτουργεί και για αυτά που δεν αποδίδουν και δεν λειτουργούν να δώσουμε συγκεκριμένε λύσεις, όχι tweet. Αυτό είναι εύκολο, το κάνω συνεχώς. Είναι πολύ πιο δύσκολο όμως να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις ως πολιτικές, ως ε, οικονομική στήριξη, προγράμματα και ούτω καθεξής. Δεύτερο, εμπορικές πολιτικές δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά δεν εγγυώνται αποτελέσματα εμπορικές πολιτικές ανοίγουν ευκαιρίες για επιχειρήσεις, εταιρείε και ούτω καθεξής και σημαντικό είναι αυτές οι ευκαιρίες να είναι με τέτοιον τρόπο που να προσφέρουν τον μέγιστο αριθμό δυνατοτήτων, στον μέγιστο αριθμό παικτών. Αυτό σημαίνει ανοιχτή εμπορική πολιτική για μένα, inclusive δηλαδή. Αυτό σημαίνει να είναι ευαίσθητη στις ανάγκες των μικρομεσών επιχειρήσεων, δηλαδή να στοχεύει στους παράγοντες που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ευάλωτες στο κόστος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα στοιχεία των εμπορικών πολιτικών που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος, αυτές θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες είναι αυτές? Για παράδειγμα, το να γνωρίζει τι γίνεται από την άλλη μεριά των συνόρων. Αυτά διευκολύνουν το εμπόριο. Η ε, ρυθμιστική δυσαναλογία. Αν έχετε πέντε διαφορετικές εμπορικές συμφωνίες με πέντε διαφορετικούς εταίρους και υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για το ίδιο προϊόν, να αυτομάτως έχετε αυτή την ρυθμιστική δυσαναλογία. Οι εμπορικές πολιτικές πρέπει να φτιαγμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν τη δημιουργία του μέγιστου αριθμού ευκαιριών για τον μέγιστο αριθμό παραγόντων. Οι εμπορικές πολιτικές όμως, είπα και πριν, δεν σας εγγυώνται τα αποτελέσματα. Εκεί μπαίνει το υπόλοιπο της ατζέντα. Τώρα για την εμπορική πολιτική συνεχίζω στα γαλλικά. Το πρόβλημα που έχετε στην Ευρώπη είναι ότι η εμπορική πολιτική είναι ομοσπονδιακή. Και ενώ οι πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης είναι εθνικές. Και σας έχει ξεφύγει η εμπορική πολιτική, την έχετε αναθέσει στις Βρυξέλλες. Ενώ οι πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης είναι εθνική υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε εσείς τον παιδαγωγικό ρόλο και τις επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επανεθνικοποιήσετε την εμπορική πολιτική, διότι αν το πράξετε αυτό, ωρεύουαρ. μπορείτε να την ξεχάσετε. Και σας ομιλώ ως πρώην διαπραγματεύτρια, ευρωπαϊκή διαπραγματεύτρια, ε. και χρειαζόμουν όλες τις χώρες μέλη ως αγορά για να με στηρίζουν απέναντι στις άλλες χώρες οι οποίες εκπροσωπούν στο κάτω γραφής χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπεται να λησμονούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές που και αυτές είναι πολιτικές αλληλεγγύης, για παράδειγμα της καινοτομίας και της έρευνας. Μεγάλη πολιτική αλληλεγγύης που επίσης κατευθύνεται από εδώ, από τις Βρυξέλλες δηλαδή. ποιος εργάζεται για τις οικονομικές πολιτικές ε, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ ο συνάδελφος του ΣΑ, γιατί εκείνοι εργάζονται πολύ για την ε, συντονισμό της παιδείας, της καινοτομίας, των συστημάτων ε, φορολόγησης, της, φορολογικής, ε, της εμπορικής πολιτικής, ε, της διεθνούς πολιτικής, ώστε να δημιουργηθεί μια πολιτική οικονομική που να είναι πιο καθολική και να περιλαμβάνει όλες αυτές τις διάφορες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάντα Κατερίνα. Εδώ βεβαίως δεν υπάρχει άμεση απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Να θυμίσουμε ότι στο επίπεδο του δίκαιου εμπορίου η ιδέα ήταν να γίνει εμπόριο υπέρ της ανάπτυξης και όχι βοήθεια να δίνεται για την ανάπτυξη. Δηλαδή, όπως είπαν πολλοί εκπρόσωποι, πολλοί ομιλητές, δεν θέλουμε τον πόρο να στηρίξει την ανάπτυξη. Ε, ποιε είναι οι δυνατότητε να αλλάξει ο ρούς της ιστορίας σε εμπορικό επίπεδο θα πρέπει να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες των πολιτών. Ε, σκέφτομαι, ας πούμε, το Fair Trade Towns υπάρχει στην Αγγλία, ε, ένα κίνημα εθελοντών που άρχισαν να συγκεντρώνονται και να οργανώνουν να σκέφτονται διαφορετικά πράγματα και υπάρχουν τώρα 1.800 fair trade και ε, σε ολόκληρο τον κόσμο και γίνεται και αυτή η πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πόλη, το βραβείο μάλλον για την Ευρωπαϊκή Πόλη του Δίκαιου Εμπορίου. Είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε όντω να λειτουργήσει ώστε να μπει το δίκαιο εμπόριο και στο συμβατικό εμπόριο. Υπάρχουν βέβαια πιέσει που μπορούν να ασχηθούν. Εμεί έχουμε μια εκστρατεία behind the prince που συζητάμε με μεγάλους ομίλους, Pepsi, Coca-Cola, τους μεγάλους ομίλους, Nestlé, Mars. Αυτές οι εταιρείες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις ιδιαίτερα όσον αφορά την ισότητα των φύλων, την, ε, την χρήση των γεών, ε, για να σταματήσει η επαλωτρίωση γεών εκεί όπου δρούν. Υπάρχει δηλαδή ένα διάλογο με αυτού του ομιλού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι καλοί και οι κακοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και αν έχουν την ευκαιρία θέλουν και εκείνοι να κάνουν κάτι το θετικό, να συμβάλλουν δηλαδή στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης εμπορικής δραστηριότητας. Επίσης ε, θα πρέπει να μπορούμε να, να, να μετρήσουμε όχι μόνο την απόδοση μιας, επί, μιας επένδυσης αλλά και τον αντίκτυπο της στην κοινωνία. Δηλαδή να έχουμε στοιχεία που μετρούν τον αντίκτυπο της κάθε δραστηριότητας στο περιβάλλον, στην ισότητα, στην ε, ισορροπία ανάμεσα στους ε, ανθρώπους και γι' αυτό υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες όμως να συνδυαστούν όσο γίνεται ε, να μην είναι ακόμα μια ανέκθεση για τις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα μια επαφή. Ε, και όσον αφορά την εταιρική ευθύνη, την κοινωνική εταιρική ευθύνη, θα πρέπει να είναι κάτι πιο αυστηρή. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει ό,τι κατεβαίνει, αλλά να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας όπως υπάρχει κώδικες διοντολογίας για τα λογιστικά ας πούμε, να μπορούμε έτσι να μετρήσουμε και τον αντίκτυπο της οικονομικής δραστηριότητας στην κοινωνία. Επίση, να δείξουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίε. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό ευκαιρίε όσον αφορά την ανάπτυξη ας πούμε, των εναλλακτικών ε, πηγών ενέργεια. Είναι μεγάλε οι ευκαιρίε για τι επιχειρήσει. Ε, ε, αλλά βεβαίω πρέπει επίση, γιατί όταν μιλάμε για προστατευτισμό, ο πρώτο που θα το υποστηρίξουν οι μεγάλοι όμιλοι που έχουν την εξουσία. Και είναι βέβαιο ότι όπως ένας πολίτης απειλείται για την ασφάλεια κτλ. Και, και μια επιτερία απειλείται όταν το επιχειρηματικό της μοντέλο απειλείται. Και εκεί θα πρέπει να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις δύσκολες κάποια στιγμή ώστε να δεχτούμε ότι κάποια επιχειρηματικά μοντέλα δεν είναι πλέον βιώσιμα στον 21ο αιώνα και για να προωθηθούν τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Και άρα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί το επιχειρηματικό μοντέλο με τους στόχους, ας πούμε, του βιώσιμη, της βιώσιμης ανάπτυξης. Να ληφθούν δεσμευτικά μέτρα, ώστε οι δραστηριότητες που έχουν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο ή υπερβελοντικό αντίκτυπο να Ε, θεωρηθούν αρνητικές και, η, το, και Τώρα, πώς ε, ε, η βιώσιμη ανάπτυξη και το δίκαιο εμπόριο θα ενταχθούν στο συμβατικό εμπόριο, κανονικά το εμπόριο θα έπρεπε να είναι δίκαιο. Το εμπόριο δημιουργεί ανάπτυξη, δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη, όπως την είδαμε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 60, ήταν μια σημαντική ανάπτυξη, ε, αλλά πρέπει επίσης να δώσουμε και μια άλλη αξία. Μια ιστορία που μου αρέσει να διηγούμε είναι Η προσφορά της δυτικής κοινωνίας είναι υπόσχεση για ένα υπέροχο εστιατόριο, όπου βλέπουμε καταπληκτικά πιάτα να σερβίρονται και όλοι θέλουμε να τα δοκιμάσουμε. Και κάποια στιγμή όταν έχουμε κάτι πια στο τραπέζι και είμαστε έτοιμοι επιτέλους να δούμε αυτό το, το πιάτο των δυτικών αξιών, μας σερβίρουν μόνο τη σάλτσα. Και βέβαια άμα δείτε τη σάλτσα στο πιάτο θα δείτε ναι είναι σάλτσα, δεν είναι το τρόφιμο. Πρέπει να έχει και πατάτες, ρύζι, κρέας, σαλάτα και αυτό ακριβώς είναι και το διακύβημα του εμπορίου, ότι κάποια στιγμή πίσω από ένα κινητό, ναι, ωραίο να έχει το κινητό, είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο, βοηθάει στην επικοινωνία, αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε μια ολόκληρη σειρά από θεμελιώδεις αξίες. Πρόεδρος Λάγκε, Ευχαριστώ βεβαίω. Καλύτερα είναι το τραπέζι πλήρε και το πιάτο σα επίση. Αλλά πράγματι καμιά φορά συμβαίνει έτσι. Κύριε Μπέρντον. Μάλιστα, οι πιο πολλέ ερωτήσει απαντήθηκαν. Αλλά έχω μια-δυο ακόμη. Ο προστατευτισμό δεν είναι νέο φαινόμενο. Το 1980 όταν άρχιζα τη σταδιοδρομία μου, η φύση τη προστασία ήταν πολύ διαφορετική, αλλά πολύ συζητιόταν τότε στην Ευρώπη ανάγκη προστασία απέναντι σε χώρε με πολύ χαμηλού μισθού. Με διάφορα εργαλεία που προτείνονταν για υφαντουργικά, για ε, ε, ρούχα και το Και μία από τις χώρες στόχους ήταν Κορέα, Νότια Κορέα, Μαλαισία, Ινδονησία. Κοιτάξτε τώρα που έχουν φτάσει αυτές οι χώρες. Εάν είχαμε τότε ε, κάνει προστατευτισμό, πού θα, πού θα ήταν αυτές οι χώρες τώρα. Η Νότια Κορέα δεν είναι τώρα τέτοια ε, ε, απειλή για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Αυτή είναι η άλλη πλευρά της, της παγκοσμιοποίησης που δεν την διηγούμαστε τόσο συχνά και που είναι αυτή που οδήγησε σε τέτοια πρόοδο. Πάντως, το επάγγελμα μου έχει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση της εμπορικής πολιτικής, ο ρόλος ανάλυσης εκεί είναι σημαντικός. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα στον τρόπο που αναλύουν το εμπόριο και τις εμπορικές πολιτικές οι οικονομολόγοι, δίνοντας υπερβολική έμφαση στις, στα κέρδη της ευημερία και λησμονώντας λίγο τις διαδικασίες, το κόστος ε, στην ευημερία των ανθρώπων και το καθεξής. Πρέπει να δούμε λίγο και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ομάδες και πώς μπορούν οι εμπορικές πολιτικές να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τις ομάδες αυτές να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση αυτή την οποία, στην οποία πρέπει να ανταποκριθούν οι οικονομολόγοι. Και βλέπουμε τώρα και μια αντίδραση από ορισμένου πολιτικού που λένε δεν χρειαζόμαστε περισσότερε αναλύσει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λάθο. Αλλά οφείλεται στον τρόπο που γίνεται η ανάλυση και στην ποιότητά τη. Δεύτερο θέμα ότι ο κόσμος είναι ε, επικριτικός απέναντι στην εμπορική πολιτική. Νομίζω ότι ο οργανισμός μου πάντως έχει και θα συνεχίσει να στέκεται κριτικά απέναντι στις εμπορικές πολιτικές όπου θεωρούμε ότι αυτές υπονομεύουν την ανάπτυξη. Έχουμε συμβάλει άλλοτε, άλλωστε στη συζήτηση σχετικά με τη CPA ε, και ιδίως για τις, ε, τους κανόνες προέλευσης και βεβαίως για τις συμφωνίες anything but arms, οτιδήποτε πλην εξοπλισμών. Εκεί όπου οι κανόνες προέλευσης είναι πολύ περιοριστικοί στον παράλληλο ε, τομέα στις αφρικανικές χώρες που ε, απασχολούν πολλές γυναίκες, ο παράλληλος τομέας δηλαδή. Αν λοιπόν ήμασταν λιγότερο περιοριστικοί στον ε, στους κανόνες προέλευσης θα, θα βλέπαμε τότε στον παράλληλο τομέα να εργάζονται περισσότερες γυναίκες στην Αφρική. Αυτό λοιπόν είναι και θα ήταν και αποτέλεσμα και μιας ε, ε, βελτιωμένης ανάλυσης. Ευχαριστώ ο πρόεδρος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ και πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους πανελίστ και τον δύο πάνελ άλλωστε, καθώς και τον κύριο Βίνκλερ που διεύθυνε μέρο τη συζητήσεως. Πραγματικά μας δώσατε μια θαυμάσια εικόνα του πού βρίσκεται το διεθνές εμπόριο. Και βεβαίω και με στόχευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με ευρύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Μας δίνεται πολύ τροφή για προβληματισμό εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Μου φαίνεται όμως επίσης σαφές ότι η εμπορική πολιτική δεν μας έπεσε από τον ουρανό. Άνθρωποι την έφτιαξαν. Και βεβαίω αποτελεί μια επιλογή και η επιλογή αυτή μπορεί και να αλλάξει και η εμπορική πολιτική και οι εμπορικές πολιτικές. Και να βάλουμε έτσι σωστά τις προτεραιότητές μας. Ίσως οι SEG να μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος μπούσουλα. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσουν την πηξίδα. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους. Και όπως είπε ο αγαπητός Βίνφλερ, ας συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ.